Um, Ο πρόεδρος Μωράης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μαθαίνω ότι πολλοί κάτω προσπαθούν να περάσουν ακόμη την ασφάλεια για να έρθουν στη συνεδρίαση. Αντιλαμβάνομαι ότι θα έρθουν και άλλοι. Αλλά προφανώς πρέπει να αρχίσουμε και αντιλαμβάνομαι βεβαίω και ότι έχετε και άλλες υποχρεώσεις, αλλά πρέπει να αρχίσουμε. Με μεγάλη μου χαρά δε, σας καλωσορίζω στην κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Θεμελιωδών Ελευθεριών και της Επιτροπής Αναφορών. Θα συμπροεδρεύσουμε εγώ και η Σεσίλια Βίξτρομ Πρόκειται για μια πραγματικά ε, στενή συνεργασία και πολύ ισχυρό συνδυασμό ε, για θέματα ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Έχουμε συζητήσει τελευταία και για τη Βρετανική αποχώρηση. Και όταν συνεργάζονται δύο κοινοβουλευτικές μας επιτροπές, η επίπτωση των εργασιών μας είναι πραγματικά πολύ σημαντική. Η σημερινή κοινή συνεδρίαση μεταξύ των δύο επιτροπών μας για την ανιθαγένεια νομίζω ότι αποτελεί ένα θετικό βήμα, διότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο χρειάζεται ανανέωση, δηλαδή χρειάζεται να συζητηθεί ξανά και ξανά. Και βεβαίως και χρειάζεται και ανάληψη δράση. Γνωρίζω ότι τέτοιες συζητήσεις γίνονται στις χώρες μέλη και στη δική μου χώρα μέλος. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από την άποψη των μέσων μαζικής επικοινωνίας για ζητήματα ανιθαγένειας, για την ανιθαγένεια παιδιών για την χορήγηση ηθαγένεια σε παιδιά και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ και τα μέλη που είναι ήδη παρόντα. Είναι πέμπτη απόγευμα, έτσι δεν είναι. Ελέγχω πάντως, ρωτώ την Σεσίλια για να μου το επιβεβαιώσει. Και οι δυο χρειάζεται να... Και η κυρία Μετσόλα γνωρίζει, η συγκήτρια. Α, είστε και, είστε και στις αναφορές κι εσείς και αντιπρόεδρος των αναφορών. Α, θαυμάσια. Ε, μιλός στην ε, κυρία Μετσόλα. Ε, Βεβαίω και οι δύο επιτροπές αυτές είναι πολύ δραστήριες, αυτό εννοούσα. Α, αν εννοείται ότι όλοι εργαζόμαστε τόσο πολύ, βεβαίω είμαστε πάντοτε απασχολημένε, ε, λέει η κυρία Βουστρόμ. Και ήθελα να απευθύνω το καλό ορίσατε στους ευρωβουλευτές που είναι παρόντες και στις ευρωβουλευτές βεβαίω η κυρία Στενόκα που είναι και ε, η συγκέντρια του Λαϊκού Κόμματος και πολύ δραστήρια στον χώρο αυτό και, και μία από τις αναφέρουσες για μία από τις χώρες που εμπλέκονται. Θα ακούσουμε λοιπόν περισσότερα από τα πρόσωπα αυτά και βεβαίως θα έρθουν και άλλοι συναδελφοί μας. Θα κάνω μια σύντομη εισαγωγή πριν να παραδώσω το μικρόφωνο στην κυρία Βίξτρομ. Ε, Μεταδίδεται από το διαδίκτυο η διαδικασία, δηλαδή τα πάντα καταχωρίζονται. Οτιδήποτε πείτε, οτιδήποτε ε, κάνετε, θα φαίνεται, ε, θα σας παρακολουθεί το κοινό και βεβαίως θα ακουστούν ό, τα όσα πείτε και πέραν των χώρων της αιθούσης. Αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα έχουν σχέση με την ανιθαγένεια. Ζήτημα βέβαια εθνικής αρμοδιότητας, όμως υπάρχει, υπάρχουν καθαρές επιπτώσεις και για το ευρωπαϊκό επίπεδο και θέτουν θέματα ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων που σαφώς είναι ζήτημα αρμοδιότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και σε θέματα ε, μετανάστευσης και ασύλου. Ασχολούνται και απασχολούνται οι συναδελφοί μου και από την Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών και από την Επιτροπή Αναφορών σχετικώς με αναφορές που τους έχουν υποβληθεί πρόσφατα. Ένα από τα πρώτα θέματα, πρώτα θέματα για την Επιτροπή Θεμελιωδών Ελευθεριών περισσότερο είναι ακολουθώντας τη λογική των συνθήκων που λέει ότι αν θα γεννεί πρόσωπα τρίτων χωρών υπό την ισχύ των, των κοινών πολιτικών Ορισμένοι ωστόσο που έρχονται δεν είναι μετανάστες, έχουν γεννηθεί εδώ και θέματα απόκτησης εθαγένειας εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ε, Ένωσης. Θα αρχίσουμε πρώτα-πρώτα με την αδυναμία των προσώπων, ε, των ανιθαγενών προσώπων να ασκήσουν τα πολιτικά τους δικαιώματα. Το Κοινοβούλιο έχει εγκύψει το θέμα αυτό κατά επανάληψη, αρχίζοντας με την κύρωση των δύο συνθήκων των Ηνωμένων Εθνών του 1954 για την Ιθαγένεια και του 1961 για την μείωση των αριθμών των ανιθαγενών. Το 2015 αναθέσαμε μελέτη σχετικά με πρακτικές και προσεγγίσεις των χωρών μελών για την αποτροπή και την λήξη της ανιθαγένειας. Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν ανάπτυξη της έκθεσης αυτής από ε, έναν ή μίαν από τους συγγραφείς της. Τώρα το Συμβούλιο έχει λάβει θέση με συμπεράσματα στα τέλη του 2015. Σήμερα λοιπόν είναι πράγματι επίκαιρη η συζήτηση αυτή σε ακρόαση. Η ακρόαση θα διαρθρωθεί σε τρία τμήματα. Πρώτα, παρουσιάσεις της καταστάσεως της χώρες μέλη για το πώς θα προληφθεί και θα πάυσει η ανιθαγένεια. Δεύτερον, μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος των ανιθαγενών παιδιών. Ε, πράγμα, θέμα πάρα πολύ ε, ε, καυτό σε πολλές ε, χώρες Τέλος, η προστασία ανιθαγενών προσώπων με τον εντοπισμό τους και την προστασία τους απέναντι σε αυθαίρετες κρατήσεις. Θα ακούσουμε και από οργανισμούς που ασχολούνται όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης, τον ΙΠΑ, το Αρμοστή των ΗΠΑ για τους Πρόσφυγες και τον Οργανισμό Θεμελιωτών Ελευθεριών. Παρούσες είναι και οργανώσεις προστασίας ανθρώπινων δικαιωμάτων, αλλά επειδή συνεργαζόμαστε σήμερα στην κοινή αυτή συνεδρίαση και με την Επιτροπή Αναφορών, θα παραδώσω με μεγάλη χαρά μετά την μακρά αυτή εισαγωγή το μικρόφωνο στην Σεσίλια Βίξτρομ, για να πει κάποια λόγια, λόγια εισαγωγικά, την οποία βεβαίω καλωσορίζω, και μετά θα συμπροεδρεύσει μαζί μου. Ευχαριστώ αγαπητέ Κλοντ, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι προσκεκλημένοι. Είναι μεγάλη η χαρά που σας ε, υποδεχόμαστε στην κοινή συνεδρίαση αυτή, όχι βεβαίως μόνο εμείς οι δύο φίλοι που βρισκόμαστε εδώ στο Προεδρείο, αλλά και όλα τα μέλη των δύο αυτών κοινοβουλευτικών επιτροπών. Έχουμε λάβει στην Επιτροπή Αναφορών μεγάλο αριθμό αναφορών για την ανιθαγένεια. Η πλέον πρόσφατη είναι αυτή που αναφέρεται σε παιδιά, σε ανιθαγενή παιδιά από εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανιθαγένειας και ε, θα τα συζητήσουμε αυτά μετά σήμερα. Το ζήτημα της ανιθαγένειας παραμένει σε υψηλή πολιτική προτεραιότητα. Η ανιθαγένεια είναι, παραμένει άλλωστε, πρόκληση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το άρθρο 15 της Παγκόσμιας Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προβλέπει ότι κάθε άτομο έχει δικαίωμα σε ηθαγένεια. Εκτός από το ότι προσβάλλεται το δικαίωμά τους αυτό, οι ανηθαγενείς αντιμετωπίζουν και πάρα πολλούς κινδύνους ε, δηλαδή ε, παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων τους. Αν ηθαγενή τέκνα ε, ενδέχεται να μεγαλώσουν χωρίς δικαιώματα, χωρίς πρόσβαση στην εκπαίδευση, χωρίς πρόσβαση σε φροντίδες υγείας και εν τέλει μένουν τα παιδιά αυτά χωρίς όραμα, χωρίς όνειρα, χωρίς ελπίδα για το μέλλον. Κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά θλιβερό. Ορισμένα ανιθαγενή παιδιά στην Ευρώπη έφτασαν κάποτε εδώ ως πρόσφυγες και ως πρόσωπα τα άσυλο. Ωστόσο, ο μεγάλος αριθμός των αληθαγενών παιδιών στην Ευρώπη γεννήθηκαν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Για αυτό το λόγο η Επιτροπή Αναφορών θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη οι χώρες μέλη της Ένωσης να αναλάβουν δράση για να προλάβουν, να αποφύγουν τα παιδιά αυτά να μεγαλώσουν χωρίς ηθαγένεια και χωρίς όνειρα για το μέλλον. Είμαι πεπισμένη ότι η σημερινή ακρόαση θα μας προσφέρει μια θαυμάσια ευκαιρία να στοχαστούμε γύρω από το θέμα αυτό και ελπίζω ότι θα μας προσφέρει και κάποιες απαντήσεις σχετικά με το πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ανιθαγένειας. Άπαξ και διαπαντός. Εύχομαι σε όλους και όλους καρποφόρα συζήτηση και χωρίς άλλη καθυστέρηση ευχαρίστως να ε, καλωσορίσω την κυρία Κάθια Σουάγκερ που έχει συντάξει την μελέτη που αναθέσαμε εμείς για λογαριασμό της ΛΥΜΠΕ για τις πρακτικές που αναλαμβάνουν οι χώρες μέλη για να ε, οδηγήσουν σε λήξη την κατάσταση αυτή της ανηθαγένειας. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή σας. Έχω πράγματι την έκθεση που συντάξαμε σήμερα μαζί με άλλους δύο συντάκτες οι οποίοι δυστυχώς κολλείονται σήμερα διότι παρακολουθούν ε, την παρουσίαση ενός διδακτορικού που γίνεται σήμερα στο Πανεπιστήμιο. Πάντως ε, θα τα πω εγώ. Και αυτό που ήθελα να πω σήμερα, ήθελα να... Αν νομίζω ότι δεν λειτουργεί το σύστημα για την ε, αλλαγή των διαφανείων. Μπορεί κάποιος να αλλάξει τις διαφάνειες. Θα παρουσιάσω σύντομα την έκθεσή μας, ένα μέρος μόνο, γιατί βεβαίως η μελέτη έχει 100 σελίδες. Έχω λοιπόν ε, ε, πάρει ένα θέμα που νομίζω ότι θα είναι ενδιαφέρον να συζητήσουμε σήμερα για το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανιθαγένεια από τώρα και ε, στο μέλλον. Θα μιλήσω και για μέτρα soft law, ήπιου δικαίου δηλαδή, ή ατελούς δικαίου, που δεν προβλέπει κυρώσεις επομένως, και ε, θα καταλήξω και συμπεράσματα τα οποία ίσως μπορέσουμε μετά να συζητήσουμε. Εξακολουθούν να μην λειτουργούν οι διαφάνειες. Έχουμε λοιπόν, τελικώς φαίνεται πως λειτουργούν. Η έκθεσή μας αποτελείται από τέσσερα τμήματα. Στο πρώτο αναφερόμαστε στα πρότυπα διεθνή και ευρωπαϊκά για την ηθαγένεια. Δεύτερο, έλεγχος κατά πόσο συμμορφώνονται με τα πρότυπα αυτά οι χώρες μέλη. Μελετούμε κάθε πρότυπο ξεχωριστά. Τι γίνεται, για παράδειγμα, για το εάν μπορεί να αφαιρεθεί η ηθαγένεια από υπόπτους για τρομοκρατία και μετά παρακολουθούμε κάθε συγκεκριμένο πρότυπο και τον τρόπο με τον οποίο συμμορφώνονται οι χώρες μέλη. Και τα έχουμε βάλει και σε πίνακες ώστε να μπορείτε να ε, λάβετε τις προφορίες αυτές πιο εύκολα. Ιδίω για την πρόληψη και της ανηθαγένειας. Μετά έχουμε στην προστασία των ανηθαγενών. Έχουμε πάρει τρεις χώρες οι οποίες έχουν διαδικασίες καθορισμού ή σχεδιάζουν να την περιλάβουν, ε, κάτω χώρες Ουγγαρία και Ενωμένο Βασίλειο. Τελευταίο μέρος, το τέταρτο, στο οποίο θα αυτό σήμερα, είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι μπορεί να κάνει στο μέλλον για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ανιθαγένειας. Ε, περί αυτού πρόκειται λοιπόν. Λοιπόν, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλούμε πρώτα-πρώτα για το ποια αφετηρία θα επιλέξουμε, διότι δεν υπάρχουν τόσα πράγματα για την ανηθαγένεια στην ε, Ευρώπη σήμερα, σε σύγκριση για παράδειγμα με το δίκαιο ασύλου. Δεν υπάρχει ακόμα δηλαδή ε, νομοθεσία του σκληρού πυρήνα ας πούμε και είναι μια πρόκληση διότι αυτό διότι δεν υπάρχουν εσωτερικά έγγραφα για να μπορέσει να βασιστεί κανείς αλλά αυτό αποτελεί ταυτόχρονα και μια ευκαιρία διότι είναι προφανής ότι κάτι πρέπει να γίνει και χρειάζεται ένα φόρουμ για να αρχίσει κανείς να σκέπτεται για στρατηγικές κατευθύνσεις που θα πρέπει να λάβει η πολιτική αυτή και είναι, βρίσκω πολύ σημαντικό ε, το στάδιο αυτό και ιδίως οι διατυπώσεις που θα χρησιμοποιηθούν οι γενικές κατευθύνσεις που θα λάβει το λεγόμενο soft law, το ήπιο δίκαιο, αν θα στοχεύσει περισσότερο στα δικαιώματα, στις μειονότητες, πώς θα πλαισιωθεί το πρόβλημα της ανηθαγένειας. Και αυτά συμβαίνουν τώρα. Μιλούμε επίσης, ένα παράδειγμα μέτρων ατελούς δικαίου είναι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ε, ε του, ε, Υπουργών για την ανηθαγένεια του 2015. Και ένα παράδειγμα είναι, ας πούμε, το γεγονός ότι σήμερα συζητούμε εδώ και ενδεχομένως να προκύψουν κάποια έγγραφα από τη συνάντησή μας αυτή. Στη μελέτη μας προτείνουμε και άλλα μέτρα soft law πολιτικής δηλαδή, που μπορούν να ληφθούν στο μέλλον για επιμέρους θέματα και όχι μόνο γενικώ περί ανηθαγένειας και προσπάθειες λύσης, μιλούμε για παράδειγμα σχετικά με την χορήγηση ηθαγένειας σε ανηθαγενή πρόσωπα. Ξεκινούμε από την ε, συνθήκη του 1954 που έχει κυρωθεί από όλα σχεδόν τα κράτη-μέλη της Ένωσης και που έχει και ένα άρθρο για την χορήγηση ηθαγένειας και λέει ότι όσο είναι δυνατόν θα γίνει προσπάθεια να επιταχύνονται οι διαδικασίες για την χορήγηση ηθαγένειας δεν έχει το άρθρο ας πούμε ένα σκληρό πυρήνα και από αυτό να απορρέουν κάποιες απαιτήσει. Δεν λέει για παράδειγμα ότι μετά από μια τριετία όπου κάποιος κατοικεί κάπου θα πρέπει να του χορηγεί τη δαγένεια ότι η αίτησή του δεν μπορεί να απορριφθεί και διάφορα τέτοια. Είναι ένα άρθρο το οποίο παροτρύνει να αναλυθούν προσπάθειες, να γίνει προσπάθεια ε, ε, ένταξης του προσώπου κ.ο.κ. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο πράγματι μπορεί να τεθεί σε φόρουμ πολιτικής και να ενθαρρύνει τις χώρες μέλη να συμμορφωθούν με την υποχρέωση αυτή όταν προκύπτει μια σχετική ευκαιρία. Επίσης προβλέπει δημιουργία πλατφορμών για την ανταλλαγή πρακτικών για το πώς προσεγγίζουν τα θέματα της ανιθαγένειας οι χώρες μέλη και το ενδεχόμενο να τους χορηγήσουν την ηθαγένεια, αριθμούς προσώπων που ε, γίνεται δεκτές οι αιτήσει τους, εάν απορριφθούν για ποιου λόγους, ποια είναι τα εμπόδια για την χορήγηση ηθαγένεια, ίσως έτσι αναφιούν κοινά προβλήματα που μπορούν να δεχθούν και κοινέ λύσει στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα παράδειγμα λοιπόν αυτό από ε, τα όσα σας είπα. Μου δίνει την επόμενη διαφάνεια. Η επόμενη διαφάνεια, πολύ σύντομα, στην ε, δικανική δράση δράση από δικαιοσύνη ε, συνήθως βασίζεται στην ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που βεβαίω δεν μπορούμε να επηρεάσουμε εμείς την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, εξαρτάται και από το τι είδου υποθέσεις ε, καλείται να επιληφθεί και, αυτά, και αποφάσεις που θα δηλαδή στο μέλλον. Υπάρχει βέβαια και η θεωρία ότι το, η νομολογία προέρχεται και από τις περιπτώσεις, από τις υποθέσεις, από τον τρόπο με τον οποίο συζητούνται, από τον ε, τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι δικηγόροι και άλλοι νομομαθείς ε, τις διάφορες αυτές υποθέσεις. Και βέβαια που βρίσκεται τώρα η νομολογία και πώς ενδέχεται να εξελιχθεί στο μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό ε, για την εξέλιξη νομολογίας όλο αυτό. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει μακρύ ιστορικό συζητήσεως και αποφάσεων για θέματα εθνικότητας. Και Βεβαίως οι χωρισμένοι έχουν την αρμοδιότητα για την χορήγηση ηθαγένεια ή για την αφαίρεσή της, αλλά οι αποφάσει θα πρέπει να λαμβάνονται με πλήρη σεβασμό του ευρωπαϊκού δικαίου. Αυτό όμως ερμηνεύεται. Δηλαδή, ο σεβασμό του ευρωπαϊκού δικαίου για θέματα ηθαγένεια ερμηνεύεται και, από, και με βάση τι αποφάσει του δικαστηρίου. Υπάρχει μια υπόθεση σχετική με την απώλεια ηθαγένειας που κατέληξε σε ηθαγένεια και η δικαστική απόφαση λέει εκεί ότι οφείλουν εκεί να ε, εφαρμόζονται διεθνή πρότυπα, πρότυπα και η αρχή της αναλογικότητας. Εφόσον απολέσει κάποιος με την ηθαγένεια μιας χώρας μέλους, μια ε, τέτοια απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί με συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό δίκαιο ή χρειάζεται κάτι άλλο. Αυτό είναι σημαντικό για την συζήτηση περί ανιθαγένειας. Δηλαδή, οι χώρες μέλη δεν μπορούν να αποφασίσουν ελεύθερα ότι αφαιρούν την ηθαγένεια κάποιου υπηκόου Η απόκτηση τώρα της ηθαγένειας, γιατί μιλεί και για αυτά η ε, νομολογία, στα πλαίσια της ανιθαγένειας, άρα ένα λογικό βήμα για την εξέλιξη της νομολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να υπάρχει μια υπόθεση που θα μας πει τι σημαίνει ο ιδιού ρηγά του EU όταν μιλούμε για απόκτηση της ευρωπαϊκής Ιθαγένειας από ένα ανιθαγενές πρόσωπο που αν δεν μπορέσει δηλαδή να αποκτήσει την Ιθαγένεια ε, μιας χώρας μέλους θα παραμείνει ανιθαγενές. Εμείς ε, σκεφτήκαμε διάφορες περιπτώσεις όπου μπορεί να διευκρινιστεί το θέμα αυτό. Αν για παράδειγμα ένα παιδί γεννηθεί στην επικράτεια μιας χώρας μέλους που προβλέπει εκ του νόμου ότι όταν γεννείται παιδί και είναι ανιθαγενές αποκτά την ηθαγένειά του, εάν το παιδί λοιπόν κατά τα τότε λαμβάνει αυτομάτως την ηθαγένειά μας, λέει η χώρα μέλος. Άρα γίνεται ηθαγενές, ηθαγενής, εάν μπορούμε να αποδείξουμε ότι αν δεν γινόταν αυτό θα η Ιθαγένε. Η Ιταλία για παράδειγμα έχει αυτή την ε, πρόβλεψη. Όμω μια φορά υπάρχει δυσκολία ότι είναι, ε, είναι δύσκολο δηλαδή να αποδειχθεί ότι σε αντίθετη περίπτωση θα παραμείνει το άτομο ανιθαγενέ. Έτσι, κατά νόμον είναι, γίνεται μεν το παιδί ε, ε αλλά λόγω ε, προβλημάτων, διοικητικών προβλημάτων μέσα στο εθνικό δίκαιο και διαδικαστικών δυσχεριών να αποδείξει ότι κατά τα άλλα θα παρέμενε ανηθαγενές, υπάρχει δυσκολία να αποκτήσει ηθαγένεια. Άλλη περίπτωση είναι κάποιος ο οποίος ε, δεν είναι εκ του νόμου ηθαγενής, έχει όμως αξίωση και είναι για την ώρα ανηθαγενής και δεν μπορεί να υποφεληθεί από την αξίωση διότι δεν εφαρμόζεται σωστά η διατάξη του νόμου, τι θα σημαίνει τότε η μη απόκτηση της ε, ηθαγένειας σε ό,τι αφορά δηλαδή την εφαρμογή της αρχής ε, της αναλογικότητας και των διατάξεων του διεθνούς δικαίου. Λέμε στην εκθεσή μας επίσης, αναφερόμαστε στο όραμα που έχουμε σχετικά με το προς τα που θα πρέπει να κινηθούν τέτοιες υποθέσεις και προς τα που θα μπορούσαν να κινηθούν ε, στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επόμενη διαφάνεια τώρα Τέλος, θέλω να μιλήσω για ενδεχόμενη νομοθετική δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανιθαγένεια. Αρχίσαμε τη συζήτηση λέγοντας ότι η υπόθεση ηθαγένειας είναι εθνική αρμοδιότητα και αυτό εμφανίζεται πάντοτε το επιχείρημα όταν συζητούμε τέτοια πράγματα και είναι σωστό πράγματι. Οι χώρες μέλη έχουν αρμοδιότητα να νομοθετούν για ζητήματα ηθαγένειας. Όμως, η αντιμετώπιση της ανιθαγένειας μέσω νομοθετικών μέτρων δεν είναι αναγκαία μέσα από την νομοθεσία περί ηθαγένειας. Αυτή είναι μια παρανόηση η οποία ξεπηδά συχνά σε τέτοιες συζητήσεις. Ηθαγένεια είναι έλλειψη ηθαγένειας. Αλλά τα ζητήματα της ανιθαγένειας δεν είναι αναγκαστικά ζητήματα που καλύπτονται από την νομοθεσία περί ηθαγένειας. Θα εξετάσω συγκεκριμένα τι μπορεί να κάνει η νομοθεσία. Να δείξω ότι η νομοθεσία περί ηθαγένειας είναι δυνατή μέσα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ε, δικαίου χωρίς να διαλύξει τα όρια των αρμοδιοτήτων. Επίσης, κάθε νηθαγενές πρόσωπο δεν είναι μετανάστης. Κάθε νηθαγενές πρόσωπο δεν είναι μετανάστης, διότι ορισμένα από τα πρόσωπα αυτά γεννήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι σωστό. Όμως, ο μετανάστης κατά τον νόμο δεν είναι αναγκαία κάποιος ο οποίος διέρχεται τα σύνορα και αυτό είναι πολύ παράξενο και δεν είναι σαφές πάντοτε, διότι μετανάστης είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι ηθαγενής. Η διάκριση που γίνεται είναι μεταξύ μεταναστών και ηθαγενών. Και η νομοθεσία περί μετανάστευσης ασχολείται με όσους δεν είναι ηθαγενείς. Πρόκειται δηλαδή για τον αποκλεισμό από την ηθαγένεια. Τα ανηθαγενή πρόσωπα είναι λοιπόν εξορισμού μετανάστες, ακόμα και αν έχουν γεννηθεί επιτόπου, διότι δεν είναι υπήκοοι τρίτων χωρών. Αυτό λέει και το άρθρο 69 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα ανηθαγενή πρόσωπα θεωρούνται μετανάστες κατά τον νομικό ορισμό στην Ένωση, άρα το ζήτημά τους είναι ζήτημα μετανάστευσης, το οποίο ωστόσο είναι ε, συντρέχουσα αρμοδιότητα μεταξύ Ένωσης και χωρών μελών. Και το καθεστώς του ανηθαγενούς προσώπου μπορεί να συζητηθεί στη βάση ενός άρθρου που αναφέρεται στο, στην ομοθεσία περί μετανάστευσης. Και αυτό μπορεί να προβλέψει τους όρους για τον χαρακτηρισμό, για το καθεστώς ενός προσώπου, πότε μια χώρα θεωρεί ένα πρόσωπο ανιθαγενές και πότε όχι και μπορεί επίσης να ασχοληθεί και με την ανιθαγένεια σε ό,τι αφορά την επιστροφή στην χώρα προελεύσεως, το οποίο δεν ρυθμίζεται για την ώρα στην Ένωση. Αυτές είναι κάποιες σκέψεις που έχουμε κάνει. Έχουμε και κάποιες συγκεκριμένες ιδέες σχετικά με το πώς μπορεί να διαμορφωθεί η νομοθεσία τι θα μπορούσε να περιλάβει ενδεχομένως μια οδηγία. Δεν θα μπω όμως σε αυτά τα πράγματα τώρα. Πόσο χρόνο έχουμε ακόμα. Πολύ σύντομα να ολοκληρώσω με κάτι που θα ήθελα να θυμηθείτε από την παρουσίασή μου είναι ότι για την ώρα υπάρχει χώρος για ανάληψη ευρωπαϊκών δράσεων για την ηθαγένεια σε διάφορα επίπεδα. Το πιο σημαντικό ενδιαφέρον και επίγον είναι να διαμορφωθούν πολιτικές μέσω μέτρων υπείου δικαίου, soft law, ξεκινώντας από τώρα για να γίνει προβληματισμός γύρω από μελλοντικέ ε, στρατηγικές. Αυτή είναι μια γενικότερη συζήτηση που πρέπει να γίνει στο υπερεθνικό επίπεδο. Πέρα αυτού, η μείωση της ανιθαγένειας είναι δυνατόν να γίνει και μέσω του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Ελέγχου, του πώς δηλαδή οι χώρες μέλη ερμηνεύουν τους κανόνες τους για την κτίση της ηθαγένεια. Και βεβαίως είναι θέμα το οποίο μπορεί να ληφθεί και νομοθετικά. Εδώ ολοκληρώνω την παρουσίασή μου. Μου ζητήθηκε βέβαια να μιλήσω και για άλλα δύο θέματα που αναφέρονται στην έκθεση την ανησυχία για το λεγόμενο pull factor, ότι μπορεί δηλαδή η ρύθμιση να γίνει παράγοντας προσέλκυσης και άλλων μεταναστών. Εμείς ε, δεν βρήκαμε στοιχεία της διαδικασίας ε, αντιμετώπισης ανηθαγένειας να είναι pull factor. Όλες οι χώρες που μας απάντησαν και που έχουν σχετικές διαδικασίες μας είπαν ότι δεν είδαν να αυξάνονται οι αριθμοί μετά από την ε, σχετική νομοθεσία. Επίση, θέλουμε και αυτό το full factor δεν σχετίζεται με την ενηθαγενή, διότι οι ανηθαγενεί παρά το ότι είναι μετανάστες, συχνά είναι κάποιοι που δεν μετακινούνται και πάρα πολύ, οπότε είναι κάποιοι των τεσάσιλο, ε, οι οποίοι εξορισμού ε, έχουν μετακινηθεί γιατί προσπαθούν να αποφύγουν κάποιο κίνδυνο, αλλά οι ανηθαγενεί συνήθω ε, είναι κολλημένοι σε ένα μέρος, δεν μετακινούνται πολύ, οπότε ε, το pull factor δεν σχετίζεται με εκείνους, παρά το ότι υπάρχουν κάποιες μελέτες που λένε ότι αυτό είναι περισσότερο μύθος παρά πραγματικότητα. Α, και κάτι άλλο που θα σας μιλήσω είναι κάποιες διαδικασίες για καλές πρακτικές, αλλά αυτά θα σας τα πούνε οι συνάδελφοι, οπότε εδώ να βάλω ε, τελεία και ευχαρίστω να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις. βλέπετε εδώ σε αυτή τη διαφάνεια τους άλλους α, συνεργάτες που μαζί μου συντάξαμε αυτήν την ε, μελέτη. Οπότε και σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε κυρία Σουάιντερ. Ναι, ήταν πολύ ενδιαφέρον όσο μας είπατε. Συγχαρητήρια και στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ και στα άλλα πανεπιστήμια που συμμετέσχουν σε αυτή τη μελέτη. Και τώρα θα πρέπει να σας παρουσιάσω τον κύριο Αντόλφο Σομαριμπάς, ο οποίος θα σας παρουσιάσει αυτή τη μελέτη. Δείχνει ο πρόεδρος το φυλάδιο αυτό, το εγχειρίδιο αυτό και λέει για αυτό το δίκτυο μετανάστευσης και την πλατφόρμα όσον αφορά την ανηθαγένεια. Α, δεν μιλήσετε με βάση αυτό το φυλάδι. Α, όχι, αλλιώς μου τα είπαν. Τέλος πάντων, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η πρόσωπα εδώ αυτή πλατφόρμα για την ανηθαγένεια και αυτή η μελέτη που έχουμε συντάξει αφορά την ανηθαγένεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, δεν έχουμε όμως αντίγραφα εδώ, αλλά μπορείτε να το βρείτε στο website της ε, πλατφόρμας μας αυτού του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τη Μετανάστευση του EMN. Όπως ε, ανέφερε η προηγούμενη ομιλήτρια, να σας μιλήσω για αυτό το δίκτυο μετανάστευσης, το οποίο συγκροτήθηκε το 2003 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, για λογαριασμό του Συμβουλίου, ούτως ώστε να καλυφθεί ανάγκη για την ανταλλαγή αξιόπιστων πληροφοριών για μετανάστευση και άσυλο και σχετικά θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε έχουμε την απόφαση 31 του 8 που μας ε, όπλησε με μια νομική βάση. Έχουμε 29 σημεία επαφής, 27 κράτη-μέλη, συν Δανία που είναι παρατηρητής και στην Ελβετία που έχει εμπλακεί, αλλά και στην Νορβηγία που είναι τακτικό μέλος. Οπότε σε ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και σε υπηρεσίες αλλά και σε εθνικά δίνουμε όλα τα δεδομένα, όλες τις πληροφορίες που είναι ε, ως στοιχεία αξιόπιστα και έχουν σχέση με την ε, μετανάστευση και το άσυλο. Okay. How we, uh, about the... Συγγνώμη για αυτή την δυσκολία αλλαγή διαφάνεια. Δεν βλέπω το Οπότε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Τη 3 η και 4 η Δεκεμβρίου του 2015 καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το δίκτυο κάνει αυτή την πλατφόρμα, τόσο ώστε να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών. Και ο στόχος είναι να μειωθούν οι ανιθαγενείς, να αναβαθμιστεί η προστασία τους και να μειωθεί ο κίνδυνος δυσμενών διακρίσεων. Αυτά επί Λουξεμβουργιανής Προεδρίας. Οπότε και είχαμε την τιμή να υλοποιήσουμε την απόφαση για την ε, πλατφόρμα. Και εκπροσωπούμε εμείς το γραφείο του Λουξεμβουργού. Οπότε όλα αυτά ε, εγκρίθηκαν τα βήματα δηλαδή υλοποίηση τη πλατφόρμα τη 11 2016 από το Διευθύνων Συμβούλιο, Steering Board. Και είπαμε στην έκθεση ότι ένα από τα εργαλεία του EMN είναι κάποια ερωτηματολόγια ad hoc και θα πρέπει να απαντήσουν τα κράτη-μέλη μέσα σε τέσσερις εβδομάδες ή λιγότερο από την υποβολή, από την διαβίβαση αυτών. Για να δούμε πώς είναι η κατάσταση με τους θα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο στόχος. Και από 25 χώρες λάβαμε απαντήσεις. Οπότε και έτσι εκπονήσαμε αυτή τη ε, μελέτη, αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να βρείτε στο website του ΕΜΕΝ. Παρουσιάσαμε εδώ το πρώτο σχετικό κείμενο στα κράτη-μέλη στην ε, μόνιμη αντιπροσωπή του Λουξεμβούργου στις 20 Δεκάτου του 2016. Οπότε εξελίχθηκε αυτή η πλατφόρμα. Οπότε και έτσι καλύπτουμε και τα κρατημέλη και διεθνή θεσμικά όργανα και με κυβερνητικέ ε, οργάνε. Επομένω, πρόκειται για συνεργασία του ΙΕΜΕΝ, τη ε, ε, αρμοστία για του πρόσφυγε του ΟΗΕ και του ΙΕΝΕΣ. Οπότε, αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα του ερωτηματολογικού. Τέσσερα κράτη-μέλη έχουν προσχωρήσει στην σύμβαση του 1954 όσον αφορά το καθεστώ που διέπει του ανιθαγένει. Και 19 κρατημέλη έχουν προσυπογράψει την συμφωνία του 61 όσον αφορά ε, την καταπολέμηση της ανιθαγένειας. Η Δε ε, την, ε, το Λουξεμβούργο μάλλον την, και η Κύπρος επικύρωσαν τη συνθήκη αλλά δεν κατέθεσαν το σχετικό έγγραφο στον ΟΗΕ. Διαπιστώσαμε επίση ότι δεν υπάρχει ομοιογένεια μεταξύ των κρατομερών όσον αφορά τι διαδικασίε με τι οποίες καθορίζεται, αποφασίζεται το καθεστώ τη ανηθαγέννης. Έχουμε τέσσερι διαφορετικέ κατηγορίε διαδικασιών, όπω είπε ήδη η συνάδελφο πριν. Γαλλία, Ενωμένο Βασίλειο και Ουγγαρία έχουν ε, κάποιες συγκεκριμένες ε, ειδικέ διαδικασίες, μετά έχουμε κάποια άλλα κράτη-μέλη που έχουν γενικές τις ή τέλο πάντων η διαδικασία καθώς μου της ενθαγένειας περικλείεται, καλύπτεται από άλλη διαδικασία για άλλο σκοπό δηλαδή. Και επίσης έχουμε και κάποιες ε, ad hoc διαδικασίες όπως η Ιρλανδία όταν έχει να κρίνει κάποια τέτοια κατάσταση ανηθαγένειας και επίσης έχουμε και κάποιες ε, ένδικες και δικαστικές διαδικασίες όπως το Βέλγιο και η Ιταλία έχουν και τα δύο. Η διαφορά είναι ότι αν, ε, το δούμε αν κάποιος είναι κάτοικος της ε, χώρας ή όχι. Ιταλία και Βέλγιο. Επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Στα περισσότερα μέλη, και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, είναι το ότι δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ αναγνώρισης του καθεστώτος του ανεθαγενούς και από την άλλη να συνδέεται αυτή η αναγνώριση με άδεια παραμονής. Το ένα λοιπόν δεν συνεπάγεται το άλλο. Και αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα. Γιατί η πρόσβαση σε κάθε όφελος, ε, παιδεία, απασχόληση, ε, γενική πνευματική και υγεία εξαρτώνται από το τι άδεια παραμονής έχει ο καθένας. Άρα εδώ έχουμε νομικό κενό. Αυτά για τους αναθεκνισμένους στα κρατη τώρα. Όπως είπε και η προηγούμενη ομιλήτρια, τα περισσότερα μέχρι ένα σημείο διευκολύνουν την απόκτηση ηθαγένειας από πλευράς των παιδιών που γεννώνται από τους ε, ανηθαγένειες. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και κάποια κενά στην νομοθεσία. Άρα κάποιοι ανήλικοι που γεννώνται ε, δεν μπορούν να αποκτήσουν την ε, πούμε κάποια σύρα η οποία φτάνει στο Λουξεμβούργο και αποκτά παιδί δεν μπορεί να πάρει την ε, ηθαγένεια για το παιδί της. Βέβαια, με τον νέο κώδικα θα γίνει αυτό, θα ρυθμιστεί στο Λουξεμβούργο, αλλά αυτό προ παρόν είναι πρόβλημα. Επίση, άλλο. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία για τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Άρα εξισώνονται οι ασυνόδευτοι ενήλικοι με τους ενήλικες. Αλλά βέβαια το πρόβλημα εδώ είναι ότι πρόκειται για τα πρόσωπα και θα έπρεπε να τύχουν άλλες μεταχείρισεις. Η επόμενη ομιλήτρια θα σας τα πει καλύτερα από μένα αυτά, αλλά το πρόβλημα που έχουμε είναι το εξής. Τώρα με το μεταναστευτικό έχουμε πολλούς μετανάστες οι οποίοι φτάνουν με κάποια παιδιά τα οποία γεννήθηκαν κατά το ταξίδι τους σε Τουρκία ή η η ή στην Ελλάδα. Οπότε το πρόβλημα ότι αυτά τα παιδιά νομικά δεν υπάρχουν. Ε, δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι σε μία από αυτές τις χώρες που προανέφερα τα παιδιά αυτά δηλώθηκαν. Να μην διαφορετική με αυτά που έλεγε η κυρία προηγουμένω, ότι δεν μετακινούνται αυτά τα πρόσωπα, γιατί μετακινούνται και τα παιδιά μαζί τους. Τώρα, ένα καλό. Το επόμενο διαφάνεια παρακαλώ. Κάτι θετικό λοιπόν. Α, όχι, όχι, όχι, αυτό το προηγούμενο. I believe uh, this flow chart demonstrate... Uh, Σε αυτό τον πίνακα από την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ. Ε, νομίζω ότι είναι θολό, αυτός είναι εγώ δεν βλέπω καλά. Γι' αυτό, αυτός ο πίνακας. Α, τώρα, τώρα. Τώρα είναι πιο καθαρή εικόνα. Τώρα ξαναθόλωσε όμως. By my of Αυτό το φτιάξαν οι συνάδελφοι. Λοιπόν, από την επαγγελματία λέει ο μιλητή, από ένα εγχειρίδιο και οποιοδήποτε δημόσιο υπάλληλο μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτό, αν δεν ξέρει τη διαδικασία. Και προσπαθούμε αυτό να το διαδώσουμε στα κρατημέλη που δεν έχουν κάποια στάνταρ διαδικασία καθορισμού και απονομή του κάθε όδου και του χαρακτηρισμού του Αγίου Οπότε έχουμε αυτή την ε, ε, η ΕΜΕΝ και η Πενταρμοστία 18 πρώτου του 17 έγινε αυτή η διάσκεψη μέσα μεταξύ αυτών των φορέων και Βέβαια το κάναμε λάθο στιγμή γιατί το κοινοβούλιο ήταν στο Στρασβούργο και δεν μπορούσατε να έρθετε και πολλοί από εσά. Αλλά έχουμε εδώ πέρα κάποια τέσσερα συμπεράσματα βασικά που παρουσιάζουν κάποιο ενδιαφέρον. Για να μπορέσουμε να καταγνωστούμε περισσότερο την ανεργαγένεια, χρειάζεται μια πρακτική προσέγγιση όσον αφορά του ε, ευάλωτου ανεργαγενεί σε κάθε κράτο μέλο. Και επομένω ε, μα προβληματίζει το πόσο ευάλωτοι είναι οι ανήλικοι, ιδίω όσον αφορά την ανεργαγένεια. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί ανήλικοι που εξαφανίζονται. Ασυνόδευτοι, ανήλικοι εξαφανίζονται από τα κράτη-μέλη. Και όπω σα είπα, καταλήξαμε στο ότι δεν υπάρχει ενιαία διαδικασία σε όλα τα κράτη-μέλη. Ούτε ξεκαθαρή διάκριση. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε τη διάκριση τη διαδικασία για τους ανεθαγενείς και τη διαδικασία για το άσυλο γιατί δεν θέλουμε η διαδικασία αναγνώριση των ενθαγενών να χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά για τους ετούντε άσυλο. Αυτό έπρεπε ξεκαθαριστεί Επομένω, και να ένα από τα θέματα τα οποία θα πρέπει να μας αποσχολήσουν Οπότε, τώρα έχουμε το προτινόμενο σχέδιο δράση που είναι το εξή. Συντονισμό με τι μη κυβερνητικέ οργανώσει και διεθνεί οργανισμού. Υπό τη αρμοστία UNICEF και έτσι να έχουμε μια διαδικασία καταστρο... ε, καταγραφής, καταγραφής και ε, επισήμανσης των ανιθαγενών ε, ευάλωτων στα κράτη-μέλη, σαν ένα πρώτο βήμα και κατόπιν να καλύψουν και όλου, όλους τους ανηθαγενείς και έτσι να εξομονηθεί κάποια η κατάσταση. Δεύτερο σημείο θα πρέπει να έχουμε μια κοινή προσέγγιση και έτσι τα κράτη-μέλη να μπορούν να εισαγάγουν κάποιες καλύτερες διαδικασίες και καθορισμού της ανεθαγήνης σε εθνικό επίπεδο. Και έτσι να έρθει αυτός ο προηγούμενος που είναι η κυρία Σουάιντερ. Η πλατφόρμα προσπαθεί να βοηθήσει την ανταλλαγή καλών πρακτικών και να διαδώσει αυτές τις μη δεσμευτικές κατευθυντήριες. Με συναντήσεις, με ό,τι, ό,τι, ό,τι υπάρχει. Όλα αυτά να είναι στη διάθεση της πλατφόρμας και έτσι να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε να εξομαλύνουμε την κατάσταση όσον αφορά τους ανεθαγενείς. Και βέβαια οι δαπάνες αυτή τη σημερινή κατάσταση είναι σημαντικές. Ε, ας πούμε πολλές φορές είναι πάρα πολύ ακριβό κάποιος να έχει δικαστική αρρωγή. Αλλού βοηθούν οι μηχανικέ οργανώσει. τόσο πάντων, όλα αυτά να τα αντιμετωπίσουμε. Τώρα, τι θα κάνουμε στο μέλλον. Όπω γνωρίζετε, η ΕΜΕΝ e έχει δύο πλατφόρμες. Το ε, REG, δηλαδή την ομάδα εμπειρογνώμων, και την πλατφόρμα για την ανηθαγένεια, οπότε έχουμε αυτού του είδους ε, ε, το, τον χώρο εργασία που τον ονομάσουμε ΆΜΗ και εκεί μπορούν να συμμετάσχουν διεθνεί οργανισμοί, μη κοινωνικές οργανώσει και η κοινωνία των πολιτών. Οπότε και έτσι θα μπορέσουμε να ανταλλάξουμε πάσα πληροφορία όσον αφορά την ανηθαγένεια. Οπότε όποιος θέλει μπορεί να μας δώσει πληροφορίες ή να λάβει από εμάς πληροφόρηση και θα συνεχίσουμε να δίνουμε τεχνική ενημέρωση στα κράτη-μέλη όσον αφορά τα θέματα της ανεθαγένειας. και το καλό με αυτό το δίκτυο είναι ότι αν κάποιος χρειάζεται βοήθεια μπορεί να την βρει από του εμπειρογνωμόνες των και θα συνεχίσουμε την οργάνωση τεχνικών διασκέψεων, ούτω ώστε να καταγράφεται η πρόοδο που έχει επιτευχθεί, και επίσης να δούμε τι είναι αυτά που πρέπει να πετύχουμε. Κάθε χρόνο να κάνουμε μια τέτοια διάσκεψη για να βλέπουμε πώς έχουν τα πράγματα και τέλος θα προσπαθούμε ε, να διαδώσουμε το θέμα, να υπάρξει συνειδητοποίηση του θέματος στα κρατημέλη, όπως κάναμε και επί Προεδρίας Μάλτας. Το είπαμε στην συνεδρίαση της και με την Εσθονική Προεδρία και με Αυστριακή και με Βουλευτική θα κάνουμε το ίδιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία με έπρεπε να αποχωρήσει, οπότε θα αναλάβω εγώ από εδώ και πέρα την Προεδρία μόνος. Να δώσουμε απευθεία το λόγο τώρα στα μέλη της ε, Επιτροπής, των δύο Επιτροπών. Έχουμε και μία πολύ ενδιαφέρουσα ε, συζήτηση στη συνέχεια για τα ανηθαγενή παιδιά. Έχετε αναφερθεί κι εσείς σε έναν βαθμό σε αυτό το ζήτημα. Το έχουμε δομήσει την όλη συζήτηση σε τέσσερα τμήματα. Ξέρουμε ότι κάποιοι έρχονται και φεύγουν. Είτε λοιπόν έχετε γενικές ερωτήσεις, είτε ερωτήσεις ειδικού ενδιαφέροντος που έχουν ορισμένοι ευρωβουλευτές, σήμερα μπορούμε να επιδείξουμε ευελιξία. Και ίσως ακόμα και να τολμήσουμε να πάρουμε απαντήσεις από συναδέλφους που δεν έχουν πάρει ακόμα το λόγο. Αυτό βέβαια είναι μια τολμηρή κίνηση από πλευρά μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά τέλος πάντων, μην τραπείτε ε, να πάρετε το λόγο, εάν δηλαδή νομίζετε ότι γνωρίζετε καλά ένα σημείο το οποίο αναφέρεται στις ερωτήσεις, απλώς πείτε το. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ωραία. Η κυρία Τσινίτση παρακαλώ έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για την ευαισθησία που δείχνετε. Γιατί δυστυχώ έχουμε διάφορε υποχρεώσει και πρέπει να υπάρχει ευελιξία. Οπότε να ευχαριστήσω του προσκεκλημένου μα ε, που μα παρουσίασαν τη δουλειά του ε, τόσο εντελεχώς και σε βάθο. Δεν έχουμε ασχοληθεί επαρκώ με το θέμα. Απαιτείται να ασχοληθούμε, να προσέξουμε. Οπότε και αυτές οι μελέτες θα πρέπει να καλύψουν και τα νομικά ζητήματα που δυστυχώς είναι πολλά. Δυστυχώς είναι πολλές οι ε, συνέπειες του να είναι κανείς γιατί δυστυχώς δεν μπορεί να απολάβει των θεμελιωδών δικαιωμάτων, μας στην παιδεία, πρόνοια κλπ. Πρόκειται για τρομερές δεσμένες διακρίσεις που υφίστανται και ιδίω ή ανήλικοι. Και είδαμε ότι σε κάποιες ε, χώρες ε, έχει ασχοληθεί η διοίκηση με το θέμα. Έχουν ληφθεί κάποια μέτρα. Στην Ιταλία έχουμε προσπαθήσει να έχουμε διοικητικές διαδικασίες και δικαστικές διαδικασίες ούτω ώστε να ε, δίνει το χαρακτηρισμό ε, του ανηθαγενούς και κατόπιν κατά περίπτωση να δίνεται η, ε, η ηθαγένεια. Ισχύει αυτό με τους ανήλικους που γεννώνται ανιθαγενείς. και έχουν προσχωρήσει στην σύμβαση του ΟΗΕ του 1961 που ασχολεί με αυτά τα θέματα. Άρα θα πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να υπάρξουν λύσεις ομοιόμορφες και ομοιογενείς σε όλα τα κράτη-μέλη. Θα αυξηθούν οι ενεθαγενές. Είναι αλήθεια ότι δεν είναι ενεθαγενείς όλοι οι μετανάστες. Αλλά, όπως είπε ο τελευταίος ομιλητής, έχουμε πάρα πολλούς ανήλικους που φτάνουν στην Ευρώπη ασυνόδευτοι. Πολλές φορές είναι βρέφη δεν ξέρουμε η ταυτότητά τους, πολλές φορές γεννώνται κατά την μετάβαση προς την Ευρώπη, ε, αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Είναι αφόρητο να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, τέτοια πρόσωπα τόσο ευάλωτα στην Ευρώπη. Και αυτά τα πρόσωπα, ενώ φυσικά και υπάρχουν, δεν υπάρχουν νομικά. Άρα, θα πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα. Θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα πέραν του μη δεσμευτικού χωρίς άμεση ισχύ soft law και να ρυθμιστεί έτσι το καθεστώς των Ιθαγενών που να ρυθμιστεί ταυτόχρονα και το θέμα της απονομής της Ιθαγένειας θα αυξηθούν οι ανηθαγενείς. Οπότε θα πρέπει ενδελεχώς να μελετήσουμε το θέμα και να καταλήξουμε σε κάποια οδηγία που να είναι ένας ελάχιστος κοινό παρονομαστής όσον αφορά τους κανόνες που θεσπίζει, αλλά που να ισχύουν οι ίδιοι να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες σε όλες τις χώρες. Είπαμε, εμείς έχουμε κάποια ρύθμιση, αλλά αλλού δεν υπάρχει. Επίσης, για πέστε μας δύο λόγια, τι γίνεται με τους ανήλικους μετανάστες, τι γίνεται με τους μετανάστες αυτούς που είναι τόσο ευάλωτοι. Μήπως θα πρέπει να υπάρξει ειδική ρύθμιση για αυτούς. Αυτοί, αυτοί οι ανήλικοι μετανάστες είναι οι πιο ανυπεράσπιστοι θα πρέπει να του δώσουμε κάποιες μίνιμουμ εγγύησεις για τα θεμελιώδη τους δικαιώματα. Ανήλικους και ιδίως τα, τα μωρά, τα παιδάκια. Άρα αυτόν μπορούν να μας πούνε οι, οι εισηγητές. Καλό και το soft law, αλλά καλύτερη η οδηγία. Ιδίως όσον αφορά τους ανήλικους. Ευχαριστούμε πολύ. Αν με επιτρέπετε να προσθέσω και εγώ ένα δικό μου ερώτημα στα όσα ανέφερε η Καταρίνα Τσινίτσι, γιατί θεωρώ ότι ε, είναι επίκαιρα εδώ. Αναφερθήκατε προηγουμένως στον ρόλο των ΜΚΟ και στην ε, νομική αρρωγή, ε, τα αντίστοιχα επίπεδα νομικής αρρωγής ε, στα επιμέρους ε, κράτη-μέλη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, υπάρχει το PRCBC, που προσπαθεί να καταχωρήσει αν θα γίνει ανηλίκου για να πολιτογραφηθούν ω Βρετανοί υπηκοοί. Θα ήθελα μόνο να επισημάνετε περισσότερο και πιο διεξοδικά τα προβλήματα της πρόσβασης στην νομική αρρωγή όχι επειδή μειώνεται γενικά, αλλά πιο συγκεκριμένα σε αυτές τις περιπτώσεις. Και πώ έχει κατάσταση συγκριτικά σε επιμέρου κρατη κράτη-μέλη για αυτέ τι κατηγορίε υποθέσεων πρέπει να χρηματοδοτηθεί η νομική αρρωγή από τις ΜΚΟ, ε, ε, πρόκειται για δωρεές, ποια είναι η γενική δομή. Είναι καλό να έχουμε μια συγκριτική ανάλυση με βάση και τις δικές σας μελέτες για να ε, γνωρίσουμε σε μεγαλύτερο βάθος την κατάσταση, γιατί ξέρουμε ότι αυτό είναι μεγάλο πρόσκομα σε ό,τι αφορά την ε, χορήγηση ηχαγένειας στους ανηλίκους. Ο κύριος Μάνκινς, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ την κυρία Σφίλτερ για την εξαιρετική μελέτη και παρουσίαση. Το ερώτημά μου αφορά αυτούς τους ε, μη υπηκόους ε, της Λετωνίας και της Εστονίας. Στην Εστονία πρόκειται για άτομα απροσδιορίστου ηθαγένειας. Έχουν γεννηθεί στην επικράτεια των ε, κρατών αυτών και έχουν ζητήσει για γενιές στη Λετωνία δεν μπορούν ε, να συμμετάσχουν σε τοπικές περιφερειακέ ή ευρωπαϊκές εκλογές. Ε, τώρα πρόκειται περίπου το 14% του πληθυσμού της χώρας μου, τη Λετωνία. Αριθμούν τα 250.000 άτομα στη Λετωνία και 52.000 στην Εστονία. Συνάδελφοι, φανταστείτε το 14% του πληθυσμού της Ρωσίας, της Κίνας ε, ή της Τουρκίας να αποκλείεται από τέτοιες διαδικασίες. Φαντάζομαι ότι τότε θα υπήρχαν πολλά ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής, της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, με ανακοινώσεις ε, όπου θα ε, απαιτούσαμε την βελτίωση της κατάστασης. Επομένως ρωτώ, γιατί θεωρείτε ότι η αρχές της Ευρωπαϊκής δρασης με ανακοινωσεις οπου θα απαιτουσαμε την βελτιωση της καταστασης Επομένω, ρωτω γιατι θεωρειτε οτι οι αρχες της ευρωπαικης ενωσης δεν αποδίδουν μεγάλη σημασία στους μη πολίτες της Λετωνίας και της Εστονίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και κυρία Τενούκο, φαντάζομαι στο ίδιο μικρό σχήματο. Μάλιστα, ευχαριστώ. Βρίσκομαι εδώ με την ιδιότητα του πλήρους μέλους ε, της Επιτροπής Αιτήσεων, αλλά τις προηγούμενες δύο θητείες τη Επιτροπή Αναφορών, αλλά στι ε, προηγούμενε δύο θητείε ε, είχε φυγεί το ζήτημα τη ανηθαγένεια από πολλέ πλευρέ. Βεβαίω, μιλώ κι εγώ για τη χώρα μου, τη Λετωνία, αλλά και για την Εστονία, με βάση αυτά που ανέφερε και ο συνάδελφο. Πρώτα απ' όλα, κάποιες γενικές ερωτήσεις ε, προς τους συναδέλφους, ε, τους ομιλητές, να σας ευχαριστήσω για τις εξαιρετικές αυτές ε, μελέτες. προς την κυρία Σφίντερ για τον ορισμό. Φαντάζομαι ότι μεγάλο πρόβλημα υπάρχει και με την ε, διαφορά ε, στους ορισμούς που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΙΕ. Στα Ηνωμένα Έθνη όλοι όσοι δεν είναι πολίτες ε, ενός κράτους αναφέρονται ως μη πολίτες, non-citizens. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρονται ως υπήκοοι τρίτων χωρών. Third country nationals. Και ο ορισμός του υπηκόου τρίτης χώρας ε, είναι περίπλοκος, γιατί και οι ανηθαγενείς και οι μη πολίτες ε, ε, πέφτουν, εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία. Και υπάρχουν μη πολίτες που εμπίπτουν μια χαρά στην κατηγορία του πολίτη. και υπάρχουν και σε ό,τι αφορά αυτά τα άτομα και αν μεταφερθούν από τη μία χώρα στην άλλη. Αλλά όλο αυτό το πρόβλημα τη ανιθαγένειας χάνεται μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση για τους ορισμούς. Μπορώ να συνεχίσω όσο θέλετε να μιλάω για αυτό το ζήτημα, αλλά τίποτα δεν αλλάζει την προσέγγιση των ε, βουλευτών εδώ. Καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε τον ορισμό των Ηνωμένων Εθνών. Μετά, για τον ορισμό της ανιθαγένειας. Και εδώ έχουμε την περίπτωση της Λετωνίας και της Εστονίας. Μπορώ να σας θέσω αυτό το ερώτημα για την παράγραφο 3.2 της έκθεσής σας, κυρία Σφίδερ. Πρόκειται για μια συγκεκριμένη περίπτωση μη πολιτών στη Λετωνία, ε, άτομα προσδιορίστου ε, ηθαγένεια στην Εστονία. Αντίστοιχα και προς τον κύριο Σαμαρίβας, 600.000 ανιθαγενείς ε, αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η περίπτωση των Λετωνών και των Εσθονών ε, εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία των 600.000 ή όχι. Συνολικά στην Λετωνία και την Εσθονία έχουμε περίπου 300.000 άτομα αυτής της, ε, αυτού του παράξενου καθεστώτος μη πολίτες και άτομα απροσδιορίστου ηθαγένειας. Το Λετωνικό Συνταγματικό ε, Δικαστήριο αναφέρει ότι δεν θεωρούνται ούτε πολίτες, ούτε ως αλλοδαπή ή ενθαγενείς, αλλά θεωρούνται ως άτομα ειδικού ε, νομικού καθεστώτος. Και αν δείτε τι λέει το Σταγματικό Δικαστήριο για το συγκεκριμένο αυτό το ειδικό νομικό καθεστώς, με τον ορισμό που δίνεται στο 3-2, ουσιαστικά είναι πολίτες ε, που δεν ε, απολάβουν ενός αριθμού ε, δικαιωμάτων. Όπως λέτε και εσείς στο σημείο 3-2. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις ε, δεύτερης ε, κατηγορίας ε, πολιτών που κατέχουν ευρωπαϊκή θαγένεια. πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση λοιπόν. Αναφέρεστε σε αυτούς τους ανθρώπους ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Και στη Λετωνία και την Αστονία. γιατί έχουν διαβατήρια αυτοί οι άνθρωποι στη Λετωνία και την Εστονία ε, συμπεριλαμβάνονται ε, στον κανονισμό περιθεωρήσεων, δικαιούνται να ταξιδέψουν. Δεν κατανοώ λοιπόν πώς μπορεί κανείς ε, να απονέμει αυτό το καθεστώς των πολιτών δεύτερης κατηγορίας σε Ευρωπαίους πολίτες. Μακάρι να την είχα αυτή την αναφορά και στη δική μου έκθεση πριν από πέντε χρόνια. Εμεί θέλαμε τότε να επεκτείνουμε την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια, αλλά δεν τα καταφέραμε. Δεν ξέρω αν έχετε καμιά πρόταση. Επίσης, ε, καταθέσατε τροπολογίες προς μια δική μου έκθεση. Δεν μπορεί κανείς να σας κατηγορήσει ότι δεν ε, προσπαθείτε με απόλυτη αποφασιστικότητα. Βλέπω ότι είναι ενέφερε καταφατικά, οπότε σίγουρα θα έχετε απαντήσει σε, αυτό το σημαντικό ζήτημα. Ξέρετε ότι είναι και μια μακραίων ιστορία. Η Τζιν Λάμπερτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη των προτέρων, γιατί όπως και άλλοι συνάδελφοι ενδέχεται να αποχωρήσω πριν από το τέλος της συνεδρίασης, δυστυχώς ορισμένες ερωτήσεις. Ίσως έχετε απαντήσει πριν φτάσω. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει αναλάβει κάποια δράση σε αυτό το τομέα και αν ναι, υπάρχουν δυνατότητες ε, κοινή ανάληψης δράσης μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της Ευρώπης. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την ε, έλλειψη πολιτικής συνοχής Κάποια κράτη-μέλη ε, προσδιορίζουν ε, ε, την ηθαγένεια κάποιου ή το καθεστώς κάποιου, λένε ότι είναι ανηθαγενής και σταματούν εκεί. Δεν δίνουν την άδεια παραμονής. Έχετε εντοπίσει κάποιο λόγο για τον οποίο συμβαίνει αυτό? είναι υπεύθυνα τα Υπουργεία που δεν συντονίζουν τη δράση τους. Μου φαίνεται απίστευτο. Αν και εντάξει, πολιτικό είμαι εδώ και χρόνια που θα πρέπει πλέον να μην εκπλήσω με τόσο από αυτά. Και με βάση αυτά που είπε η κυρία Κανίτσι για τις ε, νομοθετικές ε, δυνατότητες, έχουμε τροπολογίες για την ε, οδηγία περί διαδικασιών στο κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου. θα αντιμετωπίσουμε την ανηθαγένεια σε αυτό το αρχικό στάδιο. Προς το πρώτο μόλις αναφορά, μόνο αναφορά γίνεται. Θα δούμε αν ε, ε, μπορεί να γίνει κάτι με τις επιστροφές, γιατί και εκεί ε, κάποιοι ξεμένουν ε, στην κράτηση. Υπάρχουν άλλες νομοθετικές δραστηριότητες, ευκαιρίες όπου μπορούμε να πετύχουμε κάτι παραπάνω σε αυτό το σημείο. Ίσως υπάρχει κάτι στη τελευταία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τα παιδιά στο πλαίσιο της μετανάστευσης. Αλλά τι άλλο νομίζετε ότι μπορούμε να κάνουμε από νομοθετικής άποψης. Ναι, μπορούμε να υπερψηφίσουμε ένα ψήφισμα. Καλό θα ήταν, αλλά ακόμα καλύτερα θα ήταν να κάνουμε μια νομοθετική εργασία. Αυτό θα ήταν ακόμα πιο αποτελεσματικό. Ευχαριστώ. κυρία Πόστ. Ευχαριστώ, Κλοντ. Συγγνώμη που καθυστέρησα. Θεωρώ εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό το σημείο. Γιατί και εγώ ασχολούμαι με τα ζητήματα των Ρωμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ξέρω με βεβαιότητα ότι έχουμε πολλούς ανιθαγενείς Ρωμά και στην Ιταλία, ε, κατά συνέπεια των ε, πολέμων στη Βαλκανική Χερσόνησο. Έχουν περάσει πολλά χρόνια, οπότε τα παιδιά που γεννήθηκαν τότε γεννήθηκαν σαν ένα καθεστώς ανιθαγένειας. Και προς το παρόν δεν σημειώνεται, δεν βλέπω εγώ τουλάχιστον κάποια πρόοδο, κάποια βελτίωση στην κατάστασή τους. Όπως μιλούμε λοιπόν για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρωμά, είναι πολύ δύσκολο όταν κανείς δεν είναι πολίτης. Και μετά έχουμε τα παιδιά Ρωμά που γεννιούνται και γενιές και γενιές ανιθαγενών Ρωμά γεννιούνται στα κράτη-μέλη, αλλά επειδή δεν ε, καταχωρίζονται στο Μητρό Γεννήσεων και για διάφορους λόγους. Ε, θεωρώ ότι υπάρχει εδώ αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πρόκειται για άτομα που γεννιούνται στα κράτη-μέλη μας. Στην έκθεσή μου για την ένταξη των Ρωμά, απευθύνω έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί την κατάσταση στα κρατημέλη και να νομοθετήσει ε, σε ό,τι αφορά την ταυτοποίηση και προστασία των ατόμων των οποίων η ηθαγένεια δεν έχει αναγνωριστεί. Δεν έχουν πρόσβαση σε ταυτότητα. Δεν, δεν μπορούν να μετακινηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούν να πάνε σχολείο. Δεν έχουν δικαιώματα από τη γέννησή τους. Καλώ την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση οδηγίας για τον προσδιορισμό της ανηθαγένειας. Βλέπω το έχετε αυτό στην παράγραφο 5 του κειμένου και το στηρίζω αμέριστα γιατί θεωρώ ότι πρόκειται για ευρωπαϊκή ερμοδιότητα και ευθύνη αυτοί που γεννήθηκαν σε ένα καθεστώς τέτοιο ή ε, όσοι αναγκάστηκαν να ε, φύγουν από τις χώρες τους λόγω πολέμου. Αυτά τα παιδιά. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ε, μπορούν να ζήσουν υπό ένα ευρωπαϊκό καθεστώς με τα ανάλογα δικαιώματα. Μιλήσατε για 600.000 άτομα και μισή βρίσκονται στις χώρες της Βαλτικής. Ήμουν σε μια συνδιάσκεψη για την ανηθαγένεια στο Λουξεμβούργο και δεν υπήρχε ούτε καν αναφορά στους Ρωμά σε αυτά τα στατιστικά στοιχεία. Και γνωρίζω ότι Κάποια κρατημέλη έχουν εκατοντάδες χιλιάδες ανιθαγενών ε, χωρίς καμία αναγνώριση. Δεν ξέρω πώς έχει κατάσταση στην Ιταλία σε άλλες χώρες. Όμως υπάρχει τεράστιος αριθμός ανθρώπων που στερούνται ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων και εμείς πρέπει κάτι να κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους, ο οποίους υποτιθέτω ότι εκπροσωπούμε. Δεν έχω λοιπόν κάποιο άμεσο ερώτημα Πώς γίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μιλάει για αρμοδιότητα των κρατών μελών. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουν ούτε ευρωπαϊκά δικαιώματα, ούτε δικαιώματα των κρατών μελών. Πρέπει να λύσουμε αυτό το ζήτημα. Και με τα χαράς να ακούσω τι προτάσεις σα. Ευχαριστώ και βεβαίω μπορούν να το αναλάβουν και επόμενοι μελητέ αν υπάρχουν σχόλια. Η κυρία Βεργιά, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα και άκουσα μόνο ε, το τέλος ε, των παρεμβάσεών σας. Είναι φορτωμένο το πρόγραμμα της Πέμπτης, Πρόεδρε. Πρέπει να συγκεράσουμε πράγματα τα οποία είναι δύσκολο να συνδυάσει κανείς. Γιατί κάποιοι από εμάς να φύγουμε και σχετικά νωρίς. Εάν κατάλαβα καλά, αυτός ο αριθμός των 600.000 ανθαγενών στην επικράτηση τη Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένας αριθμό αμφιλεγόμενος. Ακόμα όμως και αν ε, κρατήσουμε ως δεδομένο αυτόν τον αριθμό, αν δείτε τους 600.000 ε, ανιθαγενείς στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια ε, σε σχέση με τα 10 εκατομμύρια ανιθαγενείς στον κόσμο, δεν έχουμε και πολλά να διδάξουμε στον υπόλοιπο κόσμο σε αυτό το ζήτημα. Εντάξει, είμαστε στο ίδιο μήκο κύματο, 0,7-0,8%. Περίπου το ποσοστό του ευρωπαϊκού πληθυσμού, 7-8% μάλλον, το ποσοστό του ευρωπαϊκού πληθυσμού σε σχέση με τον παγκόσμιο πληθυσμό. Οπότε εδώ Υπάρχει ένα σημαντικό σημείο προβληματισμού και αναζήτηση που θα πρέπει να αφορά πρώτα απ' όλα αυτού που είναι νηθαγενείς εδώ και γενιέ στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Θα ήθελα λοιπόν λίγο να επεκταθείτε λίγο περισσότερο σε αυτόν τον ε, αριθμό των 600.000 ανηθαγενών. και να απαντήσετε και την ε, συνάδελφο, γιατί προφανώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ούτε υπήκοοι ούτε ανιθαγενείς. Και αυτό έχει προεκτάσει ό,τι αφορά και την ευρωπαϊκή ηθαγένεια, γιατί η ευρωπαϊκή ηθαγένεια απορρέει και από την εθνική ηθαγένεια. Πρέπει λοιπόν να ενδιαφερθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά τα άτομα. Θα ήθελα λοιπόν να μας προβληματίσει αυτό το ζήτημα, πώς μπορούμε να βρούμε τα καλύτερα μέσα για να σημειώσουμε πρόοδο σε αυτήν την κατάσταση. Νομίζω ότι ε, πρέπει να είμαστε πιο θαραλέοι. Καλό είναι που κάνουμε τη σημερινή ακρόαση, αλλά να αναλάβουμε δράση. Κάνουμε ψηφίσματα για την ανιθαγένεια σε όλο τον κόσμο. Ας στραφούμε λίγο στην ανιθαγένεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις επιπτώσεις της και να μην μείνουμε μόνο στις επιπτώσεις των μεταναστευτικών ροών, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει πραγματικό ενδευρωπαϊκό πρόβλημα, το οποίο πρώτα απ' όλα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ και σίγουρα μετά τη σημερινή ακρόαση χρειαζόμαστε πραγματικά σημεία ανάληψης δράσης. Σίγουρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να καταρτήσει μια στρατηγική μετά από τη σημερινή ακρόαση. Σας ευχαριστώ. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ το χρονοδιάγραμμά μας. Θα συνεχίσουμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Να δώσουμε το λόγο στους δύο συναδέλφους για να απαντήσουν και μετά να αφήσετε, αφήσετε και κάτι που θα μιλήσουν για τους ανηλίκους. Μην απαντήσετε σε όλα δηλαδή. Ιδίω σε αυτό που είπε η κυρία Δανόκα και η κυρία Τσινίτσι, αυτά είναι τα κύρια και τα άλλα για τους ανηλίκους να τα αφήσετε στους επόμενους ομιλητές. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις ερωτήσεις σας. Αυτός ο αριθμός των 600.000 ε, υπάρχει στις περισσότερες από τις εκθέσεις. Όμως, συμφωνώ με τους προηγούμενους ομιλητές ότι ε, δεν είμαστε σίγουροι για το πόσοι ε, υπάρχουν στην Ευρώπη. Γι' αυτό και μία από τις πρώτες ενέργειες ε, της πλατφόρμας EMN ήταν να χαρτογραφήσει ακριβώς την κατάσταση. Όχι όμως ε, απευθυνόμενοι στα κράτη-μέλη, αξιοποιώντας τις ΜΚΟ για να ε, καταλάβουμε τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος. Γιατί δεν μπορούν τα κράτη-μέλη να πάνε στον οποιονδήποτε και πούνε ίσα είναι θα γεννήσει ή όχι. Με τη βοήθεια των ΜΚΟ, με την πλατφόρμα, θα προσπαθήσουμε να αποκομίσουμε μια εικόνα της κατάστασης και να πούμε στα κράτη-μέλη, ορίστε, αυτά είναι τα βασικά σημεία ανησυχίας. Για αυτά που είπε η κυρία Τσινίτση στην αρχή, νομίζω ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να καταγράψουμε ε, τα άτομα, αυτούς τους ανηλίκους που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη γνώμη μου, είναι εντελώς παράλογο να έχουμε παιδιά που έχουν φυσική υπόσταση, αλλά όχι νομική. Είναι σαν να μην υπάρχουν, δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο. Και προσωπικά ξέρω μια υπόθεση που πήγα στην αστυνομία και είπα, ορίστε αυτά τα δύο παιδιά πρέπει να πάνε στο σχολείο. Χρησιμοποιούμε λοιπόν ένα νόμο, το νόμο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, για να τα πάμε σχολείο. Γιατί ο δημόσιος υπάλληλο μας ζητούσε ε, πιστοποιητικό ε, από το Μητρό. Οπότε πρέπει και εμείς να τα εντοπίσουμε αυτά τα πράγματα και στην ομάδα εργασίας μας για τους λετωνούς συναδέλφους. Η ομάδα εργασίας ε, στο EMN Εκεί εκπροσωπούνται η Λετωνία και η Εστονία. Προσπαθούμε να δούμε πώς έχει η κατάσταση. Το τελευταίο, για να μην μονοπολίσω τη συζήτηση, για το κόστος. Το κόστος όλων αυτών των διαδικασιών αναφέρθηκε από μία ΜΚΟ στο Αμήνο Βασίλειο που λέει ορίστε αυτό είναι το κοστολόγιο και εμείς θα διερευνήσουμε ε, την κατάσταση περαιτέρω. Στα προηγούμενα κράτη-μέλη, οι ανήλικοι παίρνουν νομική αρρωγή εκτό από τη Λετωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Και είναι αρκετά δαπανηρέ αυτέ οι διαδικασίε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρέπει λοιπόν να απλουστεύσουμε αυτή την πρόσβαση για άτομα που ουσιαστικά δεν μπορούν καν να πιάσουν δουλειά. Και εδώ φτάνω στο τελευταίο σχόλιο μου. Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι λογικό κάποιος να πάρει το καθεστώς του ανηθαγενούς και μετά να μην έχει καμία πρόσβαση. Είχαμε μία διαβόητη υπόθεση στο Λουξεμβούργο, γιατί αυτό το άτομο πήρε το καθεστώς του ανηθαγενούς, αλλά δεν είχε δικαίωμα παραμονής. Γιατί δεν υπάρχει καμία διασύνδεση στο ε, μεταναστευτικό δίκαιο με τον ε, ορισμό του ανιθαγενούς. Έπρεπε λοιπόν να πάμε σε ανθρωπιστικό καθεστώς και περισσότερε ε, διαδικασίες που προσδιορίζουν την ανιθαγένεια προϋποθέτουν και προαπαιτούν την νόμιμη ε, διαμονή στη χώρα. Πρώτον, και αυτό είναι κάτι που εμεί εμείς ε, προάγουμε στην πλατφόρμα, έγκαιρη καταγραφή και καταχώρηση. Και το ΕΑΖΟ μπορεί να το αναλάβει το καθήκον στα hotspot και οι αρμόδιες αρχές, η Frontex, μπορούν να κάνουν αυτή την ε, αρχική καταγραφή όταν δεν έχουν ε, ε, πιστοποιητικά χαρτιά οι ανήλικοι, ιδίως οι συνόδευτοι ανήλικοι. Μετά, πρέπει να προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε μια διασύνδεση και αυτό μπορεί να γίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή, αν κάποιο παίρνει το καθεστώ ανηθαγένεια, να έχει ε, κάρτα διαμονή στη χώρα που του χορηγεί αυτό το καθεστώς. Υπό αυτή την έννοια μπορούμε λοιπόν να νομοθετήσουμε χωρίς να μπούμε στον τομέα των ε, δικαιωμάτων του πολίτη. Και για την νομική αρρωγή και το κόστος, σε κάποιες περιπτώσεις είναι απίστευτο ότι ε, το παιδί έχει το βάρος της απόδειξης. Συνήθως ε, κάποιες χώρες λένε ότι το βάρος της απόδειξης ε, ε, το επομίζεται ο ετών. Αλλά φανταστείτε ο ετών να είναι ένα παιδί. Πώς γίνεται αυτό. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα να νομοθετήσει επί αυτών των διαδικασιών και το EMN είναι κατεθειμένο να δώσει ό,τι πόρους διαθέτει για την κατάρτιση κατευθυντηριών γραμμών ή για οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο για τους διεθνείς οργανισμούς. Όπως είπα δεν είναι 600.000 ε, ο αριθμός, δεν είναι αυτός ο αριθμός που με τρομάζει μάλλον, αλλά ο τεράστιος αριθμός ε, ανηλίκων που έρχονται και δεν έχουμε καν μια εικόνα της πραγματικής κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολλά ακόμα μπορείτε να πείτε, αλλά έχουμε και άλλους εξαιρετικούς ομιλητές, οπότε μπορείτε να επανέλθετε στη συνέχεια. Κυρία Σφάιντερ, θέλετε να απαντήσετε σε κάτι συγκεκριμένο. Μάλιστα, δεν θα απαντήσω στα των ανηλίκων γιατί σίγουρα θα επανέλθουμε. Ήθελα όμως ε, να σταθώ σε μερικά ερωτήματα για την συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Νομίζω ήταν μια πολύ καλή ερώτηση αυτή. Και πραγματικά μπορεί να υπάρξει μια πολύ επικοινωνική συνεργασία, γιατί το Συμβούλιο τη Ευρώπη ε, ασχολείται ε, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα με τα ζητήματα ηθαγένεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει και σύμβαση για τα ζητήματα ηθαγένεια, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ηθαγένεια. Έχει Μεγάλη λοιπόν εμπειρογνωμοσύνη και γνώση σε αυτό το τομέα και δεν έχει τα ζητήματα αρμοδιότητας που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ και πολύ καιρό λοιπόν ασχολείται με αυτά τα ζητήματα. Δεν ξέρω πόσο, λειτουργεί αυτό από πολιτική σκοπιά, αλλά από πλευρά γνώσεων, εμπειρία, εγγράφων και εμπειρογνωμοσύνη θα είναι σίγουρα μια πολύ καλή ε, συνεργασία. Για την έλλειψη της ε, άδεια παραμονής θα ήθελα να σχολιάσω ότι οι χώρες που, οι χώρες που αυτή τη στιγμή έχουν κατάλληλες διαδικασίες καθορισμών ηθαγένειας, δίνουν επίσης και ε, το καθεστώς ε, παραμονής αναγνωρίζοντας ότι κάποιος είναι ηθαγενής. Υπάρχει μια περίπτωση να το κάνει αυτό η Ολλανδία. Ελπίζουμε να μην γίνει αυτό. Η κυβέρνηση λέει ότι ίσως να υπάρξει μια ειδική διαδικασία αναγνώρισης ανηθαγένειας που δεν οδηγεί όμως ε, αυτομάτως και στην άδεια παραμονής. Θα ήταν πραγματικά προβληματικό κάτι τέτοιο. Κατά τα άλλα, όλες οι χώρες που είπαν ότι εντάξει προσδιορίζουμε το, τη διαδικασία ανιθαγένειας, δίνουν αντίστοιχα, χορηγούν και άδεια παραμονής. Ήθελα μόνο να το επισημάνω. Τώρα για την νομοθετική δραστηριότητα είναι πιο πολιτικό το ζήτημα, αλλά από νομική άποψη υπάρχει μεγάλη ανάγκη ε, νομοθέτηση ε, νομικού πλαισίου για το ποιο είναι ανεθαγενή και ποιο όχι, με βάση και την ισχύωση νομοθεσία στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, έχουμε την οδηγία ε, περί επιστροφών, που λέει ότι ένα άτομο μπορεί να κρατηθεί για σκοπού επιστροφή μόνο αν υπάρχει εύλογη προοπτική επιστροφή. Πώς μπορεί όμως να εκτιμηθεί κάτι τέτοιο στην περίπτωση των ανθαγενών. Πόσο εύλογο είναι κανείς να θεωρεί ότι υπάρχει προοπτική επιστροφής. Τέτοιου είδους πράγματα. Έχουμε πολλά στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που χρήζουν διευκρίνηση ε, σε ό,τι αφορά τους ανεθαγενείς. Μπορούμε λοιπόν να θεωρήσουμε ότι για την ε, ε, χρηστή λειτουργία των νομικών μέτρων που ήδη ισχύουν απαιτείται λοιπόν και μια τέτοια διαδικασία. Και κάτι τελευταίο για τους ορισμούς, αν μου επιτρέπετε. Μ' αρέσει πολύ αυτό το θέμα. Ο προσδιορισμός του ανιθαγενούς σε σχέση με τους μη πολίτες στη Λετωνία και την Εστονία είναι μια ε, μακρόχρονη συζήτηση μεταξύ των διεθνών οργανισμών και της λετωνικής κυβέρνησης. Η λετωνική κυβέρνηση δεν βλέπει τους μη πολίτες ούτε ως υπηκόους ε, ούτε ως ε, ανιθαγενή. Και αυτό είναι προβληματικό γιατί το διεθνέ Δίκαιο ορίζει τον ηθαγενή ω έναν άνθρωπο που δεν έχει κάποια επικότητα. Είναι λοιπόν μια τέτοια ε, διτή διάκριση. Είτε κάποιο είναι ανιθαγενής είτε υπήκοο κάποιε χώρας. Δεν υπάρχει κάτι μεταξύ των δύο. Επομένω, δεν είναι δυνατόν για μια χώρα να πει, για ένα κράτο να πει ότι αυτή η ομάδα ούτε υπήκο είναι, είναι λίγο υπήκοοι, αλλά όχι και ακριβώ πολίτε είτε είναι υπήκοοι και Ευρωπαίοι υπήκοοι κατ' επέκταση, είτε δεν είναι και είναι μυθαγενείς. Είτε λοιπόν του συμπεριλαμβάνει ε, στον πληθυσμό της χώρας σου, είτε ε, μετά υπάγεται στο ε, διεθνές δίκαιο, δεν έχει εσύ έλεγχο για το ποιοι είναι και τι κάνουν. Δεν ξέρω ποιον βοηθάει το, και τι είναι πιο χρήσιμο και για εκείνου να του δούμε ω ενθαγενεί είτε ω υπηκόου, αλλά και σε διεθνέ επίπεδο αν έχουμε μη πολίτες που ε, εγκαθίστανται κάπου στο εξωτερικό και ε, κάνουν παιδιά για παράδειγμα στις κάτω χώρες, ας πούμε ότι ένα τέτοιο ζευγάρι για να είναι παιδί. Μπορεί και αυτό το παιδί να ε, καταγραφεί ως μη πολίτη στην Λετωνία, αλλά αυτό το παιδί ουσιαστικά είναι ανιθαγενές. Έχει κάποια δικαιώματα στη χώρα που γεννέται. Δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά, εάν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι είναι ανθαγενής αυτό ο ανήλικό, γιατί μετά δεν γίνονται δεκτοί από τη Λετωνία ω πολίτε. Βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτό το... αυτή τη μετέωρη κατάσταση. Δεν θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να προσθέσουμε άλλη μια κατηγορία. Είτε κάποιο είναι υπήκοο κάποια χώρα, είτε ανηθαγενή. Και αν ε, χαλάσουμε αυτή την εικόνα, χαλάμε και όλη την ισορροπία. Μάλιστα, λέτε, οι συνάδελφοί σας εδώ βρίσκονται ε, στην παρουσίαση διδακτορικών διατριβών και τώρα καταλαβαίνω γιατί. Είναι εξαιρετικό αυτό ο τομέα αυτό το πεδίο. Ε, δεν είναι βέβαια θετικό, αρνητικό είναι που κάποιο πρέπει να κάνει διδακτορική διατριβή σε αυτό το θέμα. Ξέρουμε ότι είναι πέμπτη, πολλοί συνάδελφοι θέλουν να φύγουν. Είναι αυτή η πέμπτη απόγευμα που μας τρομάζει όλους. Έχουμε καλέσει και τον Επίτροπο από πλευρά Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρωπινά δικαιώματα, αλλά δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. Πάμε τώρα στους επόμενους ομιλητές. Μέχρι 10 λεπτά παρακαλώ έκαστος, ίσως ε, να κάνετε μια σύνοψη, γιατί σε λίγο θα αρχίσουν να αποχωρούν και τα μέλη μας. Έτσι είναι οι πέμπτες στο Κοινοβούλιο. Παρακαλώ στα 6-7 λεπτά να μείνετε αν μπορείτε. Και μετά έτσι θα πάρετε και καλές ερωτήσεις σας. Ειλικρινά είναι καλύτερη αυτή η προσέγγιση. Λοιπόν, κύριε Κανάρης, από τη UNICEF. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ήδη έχουν υποθεί πολλά. Έτσι θα ε, διατρέξουν συντομία κάποια από τα ζητήματα και να δώσω και κάποιες ε, προκλητικές ε, ιδέες που ίσως απαντούν και σε κάποιες από τις ερωτήσεις για να βοηθήσουν την κατάσταση τώρα που είναι πέμπτη απόγευμα. Πολύ γρήγορα. Σας ευχαριστώ για τη διοργάνωση της σημερινής συνεδρίασης. καταδεικνύει και τις ε, σκληρές προσπάθειες που καταβάλλετε και σε αυτές τις επιτροπές και στο Κοινοβούλιο. Έχουμε μια δεύτερη τέτοια διοργάνωση ε, σε αυτό το ζήτημα και αυτό δείχνει πολλά. Είμαστε καθοδόν. Βέβαια, αυτέ οι συνεδριάσει από μόνο του δεν έχουν νόημα, δεν έχουν και αποτελέσματα. Πάμε λοιπόν στην επόμενη διαφάνεια. Είναι πολύ δύσκολο να το δείτε, αλλά ουσιαστικά το μόνο που σα ενδιαφέρει εδώ είναι οι ε, γαλάζιε στήλε, ο αριθμό των ανελίκων ετούν τον άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει επανέλθει το, στο θεματολόγιο. Πάντα ήταν εκεί βέβαια, δεν είναι καινούριο πρόβλημα, αλλά εδώ ίσως μπορούμε να αξιοποιήσουμε έστω και πρωτονιστικά αυτή την ευκαιρία των μεταναστών και προσφύγων που καταφτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια για να δώσουμε και πάλι έμφαση στην αντιμετώπιση του ζητήματο άπαξ και διαπαντό. Γιατί εδώ βλέπετε ότι αυξάνεται ο αριθμό των ανηλίκων μεταξύ των ετούντων άσυλων που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα στου τρει ετούντε άσυλο στην Ευρώπη είναι ανήλικο και τα τελευταία δύο χρόνια είναι πάνω από 400.000. Με πράσινο βλέπετε αυτούς που είναι απροσδιορίστου ή αγνώστου ηθαγένειας είτε ανηθαγενείς. Έχουμε το 2,5% εδώ αυτό το σημαντικό ποσοστό. Αυτό μας δείχνουν τα στοιχεία σε ό,τι αφορά ε, το μερίδιο των ανηλίκων που θεωρούνται ανιθαγενείς ή αγνώστου ηθαγένειας. Αυτό το 2,5% μπορεί να, νομίζει, να σας φαίνεται μικρό. Είναι ουσιαστικά γύρω στα 11.300 παιδιά. Αλλά είναι και πάλι υπερβολικός αυτός ο αριθμός. Θα πρέπει να είναι 0. Δεν γίνεται να έχουμε 11.000 και παραπάνω παιδιά που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρούνται ανιθαγενείς ή αγνώστοι ηθαγένειας. Και μετά αυτή η εναρμόνιση του, του ορισμού που αναφέρθηκε, ότι έχουμε διαφορετικές ερμηνείε για το τι είναι υπήκο και τι είναι ανθαγενή. Και το ανέφεραν και οι συνάδελφοι προηγουμένω. Προ το παρόν δεν έχουμε έναν ενιαίο ορισμό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και υπάρχει απόλυτη έλλειψη σαφήνεια για το τι κάνει ο καθένα όταν φτάνει ένα ανήλικο χωρί χαρτιά. Κάποιε φορέ μόνο τα ρούχα που φοράνε έχουν μαζί του σε ένα hot spot ε, που υποτίθεται ότι έχει το σκοπό της, της καταγραφής και της αναγνώρισης ε, των ευάλωτων σημείων και ανθρώπων. Όμως ακόμα και σήμερα υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις. Αυτό είναι και κάτι που αναφέρεται στην ανακοίνωση. Δεν έχουμε σαφή εντολή για τη Frontex, την ή άλλους διεθνείς οργανισμούς που βρίσκονται στα hot spots και για να ταυτοποιήσουν αλλά και να ερμηνεύσουν, να ακολουθήσουν τους, τις ίδιες ερμηνείες, τους ίδιους ορισμούς. Αυτά πρέπει να λυθούν γιατί βρίσκονται στο πεδίο αρμοδιοτήτων των ευρωπαϊκών αρχών. Να ε, δώσουμε ρητή εντολή σε Frontex, σε ASO, Eurostat, για την εναρμόνιση των κατηγοριών και να διασφαλίσουμε ότι θα καταχωρίζονται όλα τα παιδιά στην ε, σχετική κατηγορία. Η ενθαγένεια δεν είναι ζήτημα μόνο για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Και εδώ επαναρχόμαστε μάλλον δίνεται μεγαλύτερη έμφαση τώρα σε αυτό το σημείο εξαιτία τη κατάσταση. Αλλά έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό ανηλίκων ε, που βρίσκονται σε αυτή την ε, μετέωρη κατάσταση, είτε στη Λετωνία, στην Εστονία, τα παιδιά στη ε, Ρωμά, κυρίω στα Βαλκάνια που μετακινούνται πολύ. Και τελικά, όπως είπε η κυρία Λάμπερτ, ακόμα και επιστρέφονται χωρίς καμία ταυτοποίηση, είναι ανηθαγενείς. Πολλά παιδιά Ρωμά, μετά που έχω μιλήσει εγώ, έχουν φύγει από τα Βαλκάνια. Πάνε στη Δυτική Ευρώπη, επιστρέφονται, του βγάζουν ένα λεσέπασε. Πώ είναι δυνατόν να βρίσκουμε τρόπου επιστροφή αυτών των ανηλίκων, όχι όμω πολιτογράφησή του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό κενό. Εδώ βλέπετε τρία παραδείγματα μόνο, τα οποία θα ήθελα να επισημάνω. Ε, αν θέλουμε να δώσουμε σημαντική έμφαση σε τρεις μεγάλες ε, κατηγορίες ε, πολιτών ή παιδιών. Εδώ βλέπετε στην πρώτη ε, φωτογραφία τη ΣΥΜΠΑ τριών ετών. Η μητέρα της είναι Σύρια, ο πατέρας της ε, έχει πεθάνει, γεννήθηκε ε, καθοδόν, δεν είχαν κανένα τρόπο να νομοποιήσουν οι γονείς τον γάμο τους και επειδή δεν επιτρέπεται στις μητέρες να περάσουν την ηθαγένεια στα παιδιά τους, η ΣΥΜΠΑ είναι τριών ετών τώρα στη Γερμανία και ανηθαγενής. Αν δεν βρούμε λοιπόν πρακτικούς τρόπους να το λύσουμε αυτό το θέμα, θα στερηθεί το βασικό της δικαίωμα της απόκτησης ηθαγένειας και έτσι ε, θα ε, βιώνει καθημερινά ε, παραβίαση των ανθρωπινών της δικαιωμάτων σε όλη της τη ζωή. Κάτω δεξιά βλέπετε τον Μπραμ και την Ξάντρα και οι δύο έχουν γεννηθεί στις κάτω χώρες. Η μητέρα τους ήταν θύμα διακίνησης εμπορίας ανθρώπων από την Κίνα προς τις κάτω χώρες ποτέ δεν είχε καταγραφεί η ίδια στην Κίνα. Είναι και η ίδια ανεφαγενή λοιπόν και δεν έχει κανέναν τρόπο αυτή τη στιγμή να δώσει στα παιδιά της ε, την ηθαγένειά τους, γιατί έχουμε αυτά τα νομικά κενά. Γιατί πρέπει μόνη τη πρώτα να πάρει ηθαγένεια, να επιστρέψει στην Κίνα που δεν μπορεί. Ιδάλω θεωρούν τα παιδιά τη αγνώστου ηθαγένεια. Και αριστερά, ένα παράδειγμα τη έλλειψης ένταξη των Ρωμά στην κοινωνία. Έχουμε εδώ τη φωτογραφία του Μπεσίμ που είναι Αρμένιος μέσω της ε, μητέρας του. Γεννήθηκε όμως ε, στην Ελλάδα. Η μητέρα του δεν είχε ε, τα χρήματα να επιλύσει όλη αυτή τη διαδικασία. Επέστρεψε στην Ελλάδα. Τώρα έχει επιστραφεί λοιπόν ο Μπεσίμ, έχει επιστρέψει στη χώρα γέννησής του, αλλά δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί. Η ηθαγένεια δεν είναι μόνο πρόβλημα στην Ευρώπη. Είτε έχουν γεννηθεί, είτε έχουν φτάσει εδώ κτλ. Και η Ευρώπη και το Κοινοβούλιο έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει για να δώσει έμφαση στην ανηθαγένεια εκτό Ευρώπη. Το θέμα τη μετανάστευση απλώ μα αναδεικνύει την σύνδεση των δύο ζητημάτων. Εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο γεννιούνται και μεγαλώνουν χωρί ποτέ να καταγραφούν. Και ξαφνικά υπό το πρίσμα τη μετανάστευση καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι πρόβλημα. Και όχι μόνο για αυτά τα παιδιά, αλλά και για τι αρχέ επιβολή του νόμου σε κάποιε περιπτώσει. Εδώ λοιπόν έχουμε τη Μουκάσα, μια γυναίκα από την Ουγγάντα, που είχε το θάρρο να πάει στο δικαστήριο μετά το βιασμό της 13χρονης κόρης της. Αλλά δεν απονομήθηκε δικαιοσύνη γιατί δεν ήταν σε θέση να αποδείξει την ηλικία της κόρης της. Οπότε ε, απορρίφθηκε όλη η υπόθεση γιατί δεν είχε καταγραφεί το παιδί. Αυτό μας δείχνει λοιπόν ότι η ανιθαγένεια είναι μια πραγματικότητα, πολύ συγκεκριμένη κατάσταση και είναι το πρώτο και απαραίτητο βήμα προς μια ζωή παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Προχωρώ τώρα. Μπορεί να δοθεί τέλος, ναι. Για να μπορεί να γυφρεί το χάσμα όσον αφορά την δήλωση μιας γέννησης βλέπουμε ότι σε κάποια μέρη υπάρχει κάποιο μικρό χάσμα, μικρή διαφορά, κάπου στα Βαλκάνια, εκεί προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη διαδικασία της διεύνησης για ε, την μη περιτροπή στον ε, Ρωμά και εκεί βλέπετε τα παιδιά των Ρωμά που γίνονται στην Βοσνία σε σχέση με τα παιδιά των ε, εκεί υπηκών. Μιλάμε για 2-3% δηλαδή 40.000 παιδιά. Δεν είναι δυνατόν να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα ε, βέβαια μπορεί. Και στο Κωσυφοπέδιο επίση, μιλάμε πάλι για 2-3 χιλιάδε δηλαδή. Μα πάει κανεί μια, μια εβδομάδα στη χώρα, δεν γνωρίζει καν τα παιδιά ένα προ ένα. Οπότε τελικά ε, υπάρχει κάποια διαφορία στα θεσμικά όργανα και ε, είναι μία από τι ευκαιρίε που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, μια που προχωράμε τη διαδικασία τη ε, διεύρυνση και μιλάμε στο Υπουργείο Εσωτερικών, να μην μιλάμε μόνο για τα ε, θέματα τα μεταναστευτικά και εφαρμογή του δικαίου. Γιατί κάθε διάλογο για ανθρώπινα δικαιώματα, κάθε συμφωνία σύνδεση, κάθε συμφωνία επανεισδοχή και ε, το ίδιο σημαίνει και κάθε ε, σύμφωνο για την μετανάστευση. Πάνω τώρα παρακάτω. Τι να πω. Τα περισσότερα τα έχουν πει οι προηγούμενοι. Ε, θα πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες ομοιόμορφες και η ΔΕΦΚΟ η υπόθεση, η εσωτερικών υποθέσεων, να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και τρίτες χώρες να μπορέσουν να έχουν ε, τέτοιες διαδικασίες αναγνώρισης της ανηθαγένειας. Να δούμε πώς θα βρεθούν οι πόροι στα πλαίσια της ευρύτερης δέσμης μέτρων για την μετανάστευση, για την προστασία των ανηλίκων, ούτω ώστε να προστατευτούν τα δικαιώματά τους. Και τώρα τελευταίο, ε, εδώ, βλέπετε εδώ πέρα τα, τα σημεία εισόδου, ε, και η UNICEF και η Πατιαρμοστία ένωσαν τις δυνάμεις τους για ώστε να υπάρξει ένα κοινό μέτωπο για να βιστοποιήσουμε τους εταίρους μας, να προβάλλουμε το θέμα της ανηθαγένειας για να λάβει τέλος αυτό το πρόβλημα. Και είδαμε τι γίνεται σε κάποιες χώρες Ευρωπαϊκή Ένωση, Νορβηγία, Κατοχώρες, Αλβανία, Σερβία, ε, Δημοκρατία τη Μακεδονία, Κωσυφοπέδη κλπ. Και βλέπετε εδώ πέρα τι μπορεί να κάνει η κοινωνία των πολιτών μαζί με την κυβέρνηση για να λυθεί το πρόβλημα ε, τα βασικά σημεία για να αναθεώρηση του θεματολόγιου για τη μετανάστευση. είναι ευκαιρίες αυτές. Και επίσης ε, η συνολική ζήτηση που γίνεται για τη μετανάστευση, η υλοποίηση της ανακοίνωσης για του τους ε, ανήλικους, το, κοινοβούλιο που θα καλέσει να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα κρατή μέλη. Όλα αυτά είναι ευκαιρίες συγκεκριμένε και όλοι προσπαθούμε να έχουμε σωστά στατιστικά δεδομένα. Αλλιώ για θα παρακολουθήσουμε το αν σημειώνεται πρόοδος. Και τώρα κύριε Λόρα Φανβάς, θα λάβει το λόγο. Ευχαριστώ για την ευκαιρία. Εμείς ασχολούμαστε με την Ελθαγένεια παγκοσμίω και θέλω να σας πω κάποιες σκέψεις μου ε, τι κάνουμε τα τελευταία χρόνια όσον αφορά ε, τους ε, ανηλίκους, ε, ανηθαγενείς. Έχουμε τρία βασικά σημεία. Το καθένα από αυτά έχει φύγει, αλλά το θέμα είναι ε, το τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει και πώς. Όσον αφορά τώρα το τι συμβαίνει, ήδη τα είπαμε για την διάταξη, το θεματολογιό μας, είναι πολύ σημαντικό επίσης να μιλήσουμε για κάποια μέτρα θετικά πώς θα υλοποιηθούν, πώς θα μπορούν να απολάβουν ενήλικοι τα δικαιώματά τους. Τέτοια προσέγγιση πρέπει να γίνει. Ήδη ακούσαμε την Βερίνα και από άλλους το πόσο σημαντικό είναι να έχουν ηθαγένεια. Τα παιδιά να μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά του να συμμετέχουν στην κοινωνία, να έχουν όλα τα δικαιώματα που έχουν οι ανήλικοι, να έχουν κοινωνική ταυτότητα. Και είναι ηθαγένεια όμω Το κάνει τα παιδιά ευάλωτα, του φέρνει ανασφάλεια. Άρα το θέμα θα λυθεί πιο εύκολα όταν τα παιδιά είναι μικρά παρά αργότερα. Δεν μπορεί να του πει κανεί ότι όταν μεγαλώσει όλα θα είναι καλύτερα και από τα πραγματικά περιστατικά βλέπουμε ότι ισχύει και αυτό, ότι όσο μεγαλώνουν οι ενήλικοι, πιο δύσκολα ρυθμίσουμε το πρόβλημα. Για να δούμε τώρα ακριβώ ποιο είναι το πρόβλημα. Γιατί η ανηθαγένεια χτυπάει τα παιδιά και γιατί πρέπει να κάνει κάτι η Ευρώπη. Ένας από τους σημαντικούς λόγους είναι το ότι δεν υπάρχουν, δεν αρκούν ε, απαραίτητα μέτρα προφύλαξης, προστασίας και ούτως ώστε να προβλέπετε το να δίνεται η ηθαγένεια, να προβλέπετε λίγο μετά την γέννηση. Κάποια κρατημέλη έχουν κάποια μέτρα, αλλά αφορά μόνο τα παιδιά που γεννώνται στην χώρα από ανεθαγενείς γονείς. Για κάποια παιδιά λύνεται το πρόβλημα. Αυτά που δεν κληρονομούν την ηθαγένεια. Θα πρέπει να καταλάβουμε το δίκαιο των αλλοδαπών και τους άλλους λόγους γιατί δεν μπορούν οι ανήλικοι να κληρονομήσουν τους γονείς την ηθαγένεια. Θα πρέπει όμως να γίνει αναθεώρηση των σχετικών κωδικών ηθαγένειας. Θα πρέπει επίση να δούμε πώ εφαρμόζονται τα μέτρα προστασία για περισσότερα παιδιά που γίνονται στην Ευρώπη. Είναι πολύ απλό να του απονεμηθεί η ηθαγένεια. Συνήθω την από του γονεί κατά τον συνήθι τρόπο. Όμως χρειάζεται άλλη ρύθμιση για τα ανηθαγενή παιδιά. Άρα οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να γνωρίζουν τον νόμο. Και έχουμε συγκεκριμένα τεχνικά μέτρα. Θα πρέπει να ξέρουν πώς θα εφαρμόσουν τον νόμο οι αρχές, οι γονείς να ξέρουν τις διαδικασίες. Όλα αυτά χρειάζονται ενέργεια θετική για να υπάρξει αποδανεισματική προστασία. Και όπως ακούσατε από την Περίνα υπάρχουν περιπτώσεις οπότε τα παιδιά έχουν ηθαγένεια στην Ευρώπη αλλά δεν δηλαδή μπορούν να το αποδείξουν διότι δεν μπορούν να πάνε στο ληξιαρχείο, στο πιστοποιητικό γέννησης έχουν επομένω τις αποδείξεις για το γεννήθηκαν και τι έχουν την ηθαγένεια τελικά. Αυτά θα πρέπει να φροντίσουμε. Για να πούμε και κάτι που αναφέρει η κυρία Σβίτερο, Δηλαδή υπάρχουν κάποια παιδιά που γεννιόνται στην Ευρώπη και θα έπρεπε να έχουν ηθαγένεια ή γιατί υπάρχει αντίστοιχη συμφωνία, υποχρέωση του κράτους, είτε γιατί δικαιούνται σύμφωνα με το δίκαιο. Παρά δεν έχουν πάντα τις αποδείξεις. Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά αυτά μένουν ηθαγένεια και αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος με την ιδιότητα του πολίτη της Ένωσης και άρα δεν μπορούν να αποκτήσουν την ηθαγένεια. Να, το τι συμβαίνει. Τώρα, για το πώς. Το πώς συμβαίνουν αυτά, ε, είναι ξεκάθαρο. Γνωρίζουμε πώς λειτουργεί το σχετικό δίκαιο, γνωρίζουμε τις σχετικές υποχρεώσεις του κράτους μέλους, αλλά ακόμα για αν δεν έχουμε στατιστικά συγκεντρωτικά στοιχεία είναι σαφές τι πρέπει να κάνουμε. Τουλάχιστον όσον αφορά τα αν παιδιά. Και ένα σημαντικό μέσο είναι η συμφωνία του ε, εξενερή καταπολέμηση της ανεθαγένειας. Είναι σημαντικό να προσχωρήσουν όλα τα κρατή μέλη γιατί έχουμε εννέα τέτοια κρατή μέλη που ακόμη δεν έχουν προσυπογράψει αυτή την σύμβαση του 61. Αυτό θα πρέπει να διορθωθεί. Πέντε από αυτά τα κρατημέλη πάντως έχουν μέτρα προφύλαξης και προστασίας από την ανιθαγένεια. Οπότε πρέπει να προσυπογράψουν όλα τα κράτη την σύμβαση να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Επίσης, όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης έχουν την υποχρέωση να αναγνωρίσουν την δικαίωμα των υλίκων μέσω των διεθνών συμφωνιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών. Άρα, τα κρατημέλη έχουν θετική υποχρέωση να υλοποιούν και να σέβονται αυτά τα δικαιώματα των ανηλίκων. Ακόμα και βάσει των γενικών αρχών προστασίας αυτών. Καλύτερα, δηλαδή εξπρόσεις του συμφέροντος του παιδιού, και έχουμε την Επιτροπή του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, την υπατιαρμοστία δηλαδή, που έχει αποφανθεί όσον αφορά την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Και 16 από τα 28 κρατημέλη ήδη έχουν λάβει από αυτή την Επιτροπή του ΟΗΕ κάποιες συστάσεις για το πρόβλημα. Και πολλές φορές αυτή η Επιτροπή των Δικαιωμάτων των Παιδιών έχει διατυπώσει προτάσεις. Τσεχία, Εστονία, Ιταλία, κάτω χώρες έχουν κάποιες σχετικές διατάξεις στο δικαιό τους. Άρα θα πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν δεσμευτικές διατάξεις υπέρ των ανηλίκων και των δικαιωμάτων τους. Το πώς γίνονται τώρα όλα αυτά, πώς το πρόβλημα... Ε, μπορεί να αντιμετωπιστεί, να δούμε τι γίνεται με τους στόχους τους αναπτυξιακούς, να υπάρχει καταχώρηση σε ληξιαρχείο όλων, να υπάρχει τέτοια υποχρέωση διεθνώς πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδατε και αυτές τις μελέτες, επισημάθηκαν ποιες είναι καλές πρακτικές και έχει κάνει εκστρατεία ο ΙΕ για να καταλάβουμε καλύτερα το γιατί πρέπει με πρόληψη να αντιμετωπίζεται η ανηθαγένεια. Τέλος, έχουμε για το γιατί συμβαίνει αυτό, και πράγματα να πούμε. Υπάρχει κίνδυνο τον έχουμε όλα ένα και περισσότερα παιδιά γίνει στην Ένωση. ιδίω ως απόρρια του μεταναστευτικού. Και επίσης είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι λένε και περισσότερο προσέχουμε το πρόβλημα και αυτό φέρνει διεθνή κινητοποίηση. Και αυτό θα πρέπει να συνεπάγεται περισσότερη συμμετοχή και προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΙΕΝΕΣ ε, έχει κάνει εκστρατεία, ο ΙΕ, ε, ο συνασπισμός φορέων που είπε η και άλλες πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί. Όμως, Πέραν αυτών των πρωτοβουλειών και αυτή τη θετική τάση που πρέπει να εκμεταλλευτούμε, θα πρέπει να προσέξουμε τον κίνδυνο αύξηση των ανιθαγενών μέσω του μεταναστευτικού. Δεν θα τα ξαναπώ, αλλά να σας πω και κάτι άλλο, το οποίο είναι θέμα που εξελίσσεται και παροξύνεται. Τι γίνεται με τους Τούρκους υπηκός εκτός Τουρκίας. Πολλές φορές υφίστανται αφαίρεση της ταγενείας τους. Και η αιτία είναι το αποτυχημένο πραξιόβημα πέρσι. Μέσα σε τρει μέρε είχαμε κάποιε χιλιάδε στην και αυτό δεν μπορούσαν να το κάνουν. Εάν δεν το κάνουν, εάν δεν επανέλθουν, τότε η κυβέρνηση θα του αφαιρέσει την ηθαγένεια. Πέρσι έχουμε όλο ένα και περισσότερα περιστατικά ε, Τούρκων που δεν τους παρέχονται προξενικές υπηρεσίες, τους αρνούνται τα προξενία. Ε, τέσσερις, πρόσφατα 800 τέτοιες συνολικά και 76 τέτοιες περιπτώσεις έχουν να κάνουν με το ότι δεν τους δίνουν ε, διαβατήριο, δεν τους δίνουν επίσης και ταυτότητα για τα παιδιά τα οποία γεννούν αυτοί οι Τουρκοί υπήκοοι. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ε, άρα θα πρέπει στα σοβαρά να λάβει κάποια μέτρα να ασχοληθεί στα σοβαρά Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος Μωράης, ευχαριστώ έχετε πάντα υπόψη σας ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να αποχωρούν τα μέλη μας. Όσο πιο σύντομα η παρουσίασή σας τόσο καλύτερα γιατί θα έχουν την ευκαιρία μετά τα μέλη μας, δηλαδή οι βουλευτές, να σας υποβάλουν ερωτήσεις. Θα ακολουθήσει η Μάργαρετ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει τον ρόλο της συντονίστριας στην ε, μονάδα για ε, στην Διεύθυνση μάλλον ε, που ασχολείται με τα ε, θεμελιώδη δικαιώματα. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πραγματικά όσο γίνεται συντομότερη. Για το Συμβούλιο της Ευρώπης, στις 19 Μαΐου το Συμβούλιο της Ευρώπης ενέκρινε σχέδιο δράσεως για την προστασία παιδιών μεταναστών. Θα ιδρύσουν ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα επιβαλλει προτασεις προτάσεις 2018-19. Έχω να θέσω υπόψη σας μια περίπτωση από το Δεκέμβριο του 2016 της Ιρλανδίας σχετικά με ένα ασυνόδευτο ανιθαγενές παιδί, του οποίου υπόθεση χρειάστηκε 6 χρόνια για να λυθεί και 12 χρόνια μετά την άφηξή του στην Ιρλανδία. Η υπόθεση αυτή κατέδειξε ότι υπάρχουν διατάξεις για παιδιά ανθαγενή που γεννιούνται στην Ιρλανδία, αλλά όχι για παιδιά που μετακινούνται στην Ιρλανδία. Πολύ σημαντικό είναι και το ζήτημα των διακριτικών εξουσιών. Η υπόθεση επίσης της διαφορετικής μεταχείρισης διδήμων υπό τις ίδιες συνθήκες είναι ε, πολύ ενδιαφέρουσα. Έχουμε τώρα μία μικρή μελέτη που πρόκειται να ξεκινήσει για να καταγράψει την έρευνα για τα δικαιώματα των παιδιών Ρωμά και η ανιθαγένεια θα είναι ένα από τα θέματα που θα καλύψει και στις χώρες μέλη αλλά και χώρες της διεύρυνσης. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 12ης Απριλίου φέτος, αναφέρθηκε ήδη από άλλους ομιλητές, προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη και το ζήτημα της ανιθαγένειας σε συνεργασία και με άλλους διεθνείς οργανισμούς όπως τον είπα το αρμοστή για τους ε, πρόσφυγες των ΗΠΑ και έγινε και η παρουσίαση για τα δικαιώματα των παιδιών με πρακτικά μέτρα για την επιτάχυνση των διαδικασιών αναγνώρισης. Παιδιά που βρίσκονται σε μετανάστευση θα πρέπει πάντοτε να μπορούν να εντοπίζονται και να αναγνωρίζονται, να μπορεί να διαπιστωθεί αν ένα παιδί είναι ασυνόδευτο, έχει χωριστεί από την οικογένειά του, αν είναι άπατρη, επίσης και τα παιδιά αυτά που δεν έχουν πάντα καταχωριστεί πρέπει να καταχωρίζονται και τα άλλα τους ε, ε, στοιχεία για παιδιά που στερούνται ηθαγένειας. Εκεί πρέπει να καταχωρίζονται και ζητήματα όπως ε, το φύλλο για την ε, κατάλληλη υποδοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς μιλούμε για την ανάγκη να τους προσφερθεί εκπαίδευση, φροντίδα υγείας ανεξαρτήτως από τη χώρα στην οποία καταλήγουν, αναφερόμαστε και σε διαδικασίες καθορισμού του καθεστώτος που θα πρέπει να δοθεί στις διαδικασίες αυτές προτεραιότητα. Το ζήτημα της κυδαιμονίας ασυνόδευτων παιδιών επίσης και αυτό θα βασιστεί σε ένα δίκτυο το οποίο ιδρύεται τώρα για την κυδαιμονία ασυνόδευτων παιδιών. Σε ό,τι αφορά λύσεις με διάρκεια, βιώσιμες λύσεις, ενθαρρύνουμε τις χώρες μέλη να διασφαλίσουν την ύπαρξη διαδικασιών καθορισμού του καθεστώτος των παιδιών για παιδιά τα οποία δεν θα επιστραφούν ιδίως και ιδίω για τα παιδιά τα οποία έχουν διαμείνει στη συγκεκριμένη χώρα για κάποιο διάστημα. Και βεβαίως παρακολουθούμε όλες τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των διαφόρων οργανισμών και τι συστάσεις που γίνονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, έχουμε σήμερα κλείσιμο προτάσεων για την φροντίδα των παιδιών αυτών και ορισμένες προτάσεις, είπαμε ρητά, ότι θα καλύπτονται και υπηκοητή των χωρών και ασυνόδευτα παιδιά και ανηθαγενή παιδιά. Και λέμε επίσης ότι για τον καθορισμό της, του καθεστώτος αυτό θα πρέπει να γίνεται διαρκώς και ως ρουτίνα, διότι γνωρίζουμε ότι συχνά ότι όταν παιδιά βρίσκονται σε μια χώρα, συχνά δεν γίνεται απολύτως τίποτα για τον καθορισμό του καθεστώτος τους. περιλαμβάνουμε και ένα τμήμα στη βιβλιογραφία για, ε, το καθημερινό του καθεστώτος. Και τέλος, γίνονται προσπάθειες για να βελτιωθεί η ορατότητα των παιδιών αυτών και ελπίζω ότι σύντομα θα μπορέσουν να προκύψουν αποτελέσματα. Ευχαριστώ πολύ Μάργαρετ. προχωρήσουμε τώρα, όπως, είπατε, όπως γνωρίζετε είναι κοινή συνεδρίαση Έχουμε την αναφορά Chris Nash 0076 κάθετος 17. Θα μιλήσει βεβαίως ως αναφερόμενος, αλλά και είναι και ταυτόχρονα και εμπειρογνώμων. Αναφορά του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανιθαγένειας. και ζητεί από τις ε, ευρωπαϊκές χώρες μέλη να καλύψουν τα κενά στο δίκαιό τους, να ε, συμμετάσχουν στους διεθνείς οργανισμούς και να προβλέψουν τις σχετικές προστασίες. Και λέει ότι η Ιθαγένεια θα πρέπει να χορηγείται σε παιδιά τα οποία διαβιούν στην επικράτεια των χωρών αυτών, εφόσον υπό, εάν δεν συμβεί αυτό θα παραμείνουν η Δεν ξέρω γιατί τα λέω όλα αυτά, αφού αναμένω ότι ο ίδιος ο κύριος Κρίθνας θα τα πει όλα αυτά τα πράγματα, δεν είναι. Και εδώ μεταξύ σας ζητώ και από όλους βεβαίως να είστε σύντομοι και ασφαλώς θα τα πείτε εσείς καλύτερα από εμένα. Έχετε μάλιστα και ένα βίντεο έτσι δεν είναι. Ευχαριστώ Κρίς, μπορείτε να μιλήσετε. Είχα σκοπό ε, να κάνω προσπάθεια να συντομεύσω. Θα δείξω αμέσως και το ε, βίντεο μας. Εδώ εκπροσωπώ όχι μόνο την οργανωσή μου, που έχουμε 110 μέλη σε 40 χώρες, αλλά και τα πρόσωπα τα οποία έχουν συνυπογράψει την αναφορά μας που ζητούν από τις ευρωπαϊκές ηγεσίε να προστατεύσουν τα νηθαγενή παιδιά. Αρχίσαμε την εκστρατεία μας από το 2015, ποτέ δεν περιμέναμε τέτοια ανταπόκριση και αυτό μαρτυρεί για το γεγονός ότι το κοινό ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το θέμα αυτό. Δεν θα σας διαβάσω το κείμενο της αναφοράς, Κύριε Πρόεδρε, πολύ καλά το εξηγήσατε εσείς. Θα μιλήσω μόνο για τους λόγους για τους οποίους ξεκινήσαμε με την αναφορά. Στην βάση της έρευνας που κάναμε από το 2015 και μετά που λέμε κανένα παιδί δεν θα πρέπει να παραμένει ανιθαγενές, είδαμε ότι οι μισές ευρωπαϊκές χώρες μέλη δεν λαμβάνουν υπόψη περιπτώσεις παιδιών που γεννιούνται απάτριδα στις ε, ε, επικρατείες τους και ζητούμε να ληφθούν τρία μέτρα. Πρώτον, χρειάζεται περισσότεροι φορείς και χώρες να αναγνωρίσουν το πρόβλημα και ευτυχώς η σημερινή συνάντηση εξυπηρετεί το σκοπό αυτό. Δεύτερον, το, η λύση είναι απλή. Χρειάζονται νομοθετικές αλλαγές που δεν κοστίζουν και πολλά και ούτε άλλωστε παρεμβαίνουν στην εθνική κυριαρχία. Και τρίτο, χρειαζόμαστε εφαρμογή στην πράξη. Και εδώ ερχόμαστε σε ορισμένα από τα σημεία που είπαν οι προηγούμενες ομιλήτριες, Παλώνα Βερένα και Μάγκαρετ, το βασικό είναι η αναγνώριση, ο εντοπισμός. Εάν δηλαδή οι άνθρωποι που φτάνουν, οι γονείς των παιδιών αυτών, είναι ήδη ανηθαγενείς ή δεν μπορούν να μεταδώσουν την ηθαγένεια στα παιδιά τους. Και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και τα παιδιά τα οποία είναι ανηθαγενή και βρίσκονται στο επίκεντρο τη συζητήσεω αυτή, να μου επιτρέψετε να σα δείξω ένα σύντομο φιλμ τώρα με συμμετοχή ορισμένων από τα παιδιά που είδαμε στην έρευνά μα.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 I think the, uh, story... Πρόκειται για την ιστορία του Έρικ, της Μαρίας και του Ανδρέα που δείχνουν ποια είναι τα προβλήματα των παιδιών που μεγαλώνουν χωρίς ε, εθνικότητα και επομένως στερούνται τα δικαιώματα και την δυνατότητα να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους. Κανένα παιδί δεν επιλέγει να ε, παραμείνει ανηθαγενές, ούτε είναι ποτέ δική του ευθύνη, ούτε άλλωστε εξυπηρετεί το συμφέρον του. Ο ίδιος ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων δεν περιλαμβάνει, ε, μάλλον στο άρθρο 24 λέει ότι καλεί μάλλον τις χώρες μέλη να λάβουν μέτρα για την εξυπηρέτηση του, ε, του συμφέροντος των παιδιών. Και γι' αυτό νομίζω ότι και το Intergroup του Κοινοβουλίου για τα Δικαιώματα του Παιδιού έχει δείξει ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Έχουμε κάνει άλλε τρει συναντήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την διακομματική αυτή ομάδα Ευρωβουλευτών και θεωρώ ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ε, προσπάθεια να γίνει ένα βήμα προς τα εμπρός και να δούμε πώς μπορούμε να αναλάβουμε δράση, διότι το, την οφείλουμε την δράση αυτή στα παιδιά και όχι μόνο στα παιδιά του φιλμ, αλλά σε όλα τα παιδιά που είναι ανιθαγενείς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Προτιμώ να σταματήσω εδώ ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί η συζήτηση με τις παρούσες ευρωβουλεύτριες και ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ε, όλους τους ομιλητές, λέει ο πρόεδρος Μωράης. Έχουμε άλλους δύο ομιλητές. Θέλετε όμως εσείς να κάνετε μια σύντομη παρέμβαση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση για την κατάσταση στη Λετωνία. Είπαμε ότι έχει έρθει η ώρα να δοθεί η ηθαγένεια στα νεογέννητα παιδιά των ανηθαγενών. Θετικό μήνυμα, αλλά εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξο. Γιατί πρόκειται για θέμα υλοποίηση των καλών προθέσεων. Εγώ είμαι πρώην δημοσιογράφος και από ό,τι θυμούμε ε, έχουμε εδώ τώρα τον τέταρτο πρόεδρο της Λετωνία που κάνει τη σχετική ανακοίνωση και που τίποτε δεν γίνεται. Το 1995 στη Λετωνία το Εθνικό Κοινοβούλιο ενέκρινε νόμο για το καθεστώς προσώπων που δεν είναι ε, πλέον ε, δεν είναι μάλλον ε, πολίτες της Λετωνίας. Δηλαδή είναι non-citizens. Η Σοβιετική Ένωση κατέρευσε προ 25 ετών. Όμως οι άνθρωποι αυτοί έχουν καθεστώς πρώην πολιτών της Σοβιετικής Ένωσης και υπάρχουν παραπάνω από 6.000 παιδιά των οποίων το καθεστώς τώρα ζουν τα πρόσωπα αυτά στην Λετωνία και είναι άγνωστο το καθεστώς τους. Ερώτηση τι μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αλλάξει η κατάσταση για τα νεογέννητα παιδιά των μη πολιτών που διαβιούν στη Λετωνία. Ποιος θα επιθυμούσε να απαντήσει. Αυτό βέβαια εντάσσεται περισσότερο στα συμπεράσματα που μπορεί να προκύψουν από την συζήτηση. Είπε και η κυρία Σδανόκα ότι είναι ένα θέμα το οποίο χρονολογείται από μακρού. Θέλετε λοιπόν κάποιο εξημών να απαντήσει τώρα ή... Μήπως προτιμάτε να ακούσουμε τους άλλους δύο, γιατί έχουμε ακόμα και για την ταυτοποίηση και προστασία των ανιθαγενών. Αντιλαμβάνομαι βεβαίω ότι είναι αυτή η τρομερή υπόθεση τη πέμπτη. Οι άνθρωποι εδώ πρέπει να προλάβουν αεροπλάνα, τρένα κλπ. Διότι αλλιώ ε, αναγκαστικά θα περιμένουν μέχρι αύριο. Μπορούμε λοιπόν, ε, κύριε συνάδελφοι, αν συμφωνείτε, να ακούσουμε τους επόμενους ομιλητές και ίσως μπορούμε να καταλήξουμε στο τέλο σε κάποια συμπεράσματα. δώσουμε το λόγο λοιπόν στη Μελλοντικάνα από την υπατερμοστία του για τους Παρακαλώ να μείνετε στα 6-7 λεπτά. Ε, καλώς ήρθατε βεβαίως. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εξ ονόματο τη Υπότιτλη Αρμοσία του ΙΕ για του πρόσφυγε, θέλω να ευχαριστήσω και, τους δύο, ε, και τι δύο επιτροπέ για την δυνατότητα ε, που μου δίνουν να μιλήσω σήμερα σε αυτή τη σημαντική ακρόαση. Θα προσπαθήσω να τηρήσω το χρονικό όριο που θέσατε. Τα Οι γραπτέ μου παρατηρήσει ήταν γύρω στα 10 λεπτά. Κάποια ζητήματα έχουν ήδη απαντηθεί από άλλου συναδέλφου. Θα προσπαθήσω λοιπόν να διατρέψω συντομία κάποια σημεία, να προσθέσω και να συμπληρώσω σε κάποια άλλα και να καταλήξω σε κάποιε συγκεκριμένε ε, συστάσει προ την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κρατημέλη. Πρώτον, δεν θα γνωρίζετε, το 2014 η αρμοστία του ΙΕ για τους πρόσφυγες ξεκίνησε μια πολύ φιλόδοξη εκστρατεία να σταματήσει, να δοθεί ένα τέλος στην ανηθαγένεια μέχρι το 2024 και είναι πολύ σημαντικό για μας που ε, σημειώνεται και δίνεται σημασία σε αυτό το θέμα και ήδη ενθαρρύνεται τα κράτη-μέλη να αναλάβουν δράση για την ανηθαγένεια μέσω μιας σειράς ψηφισμάτων και εκθέσεων. Με τα χαρά σας ήθελα να ανακοινώσω ότι στο δεύτερο εξάμεινο του 2019 ε, είπατε αρμοστέτο για τις πρόσφυγες, θα διοργανώσει μια εκδήλωση υψηλού επίπεδου ε, για την ανηθαγένεια στα μισά ακριβώ εκστρατεία και ε, περιμένουμε και την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Κρατών Μελών για να και με την προσέλευσή τους αλλά και με υποσχέσεις να κάνουν περισσότερα και μέσω της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παροτρύνουν και άλλους ε, να παρευρεθούν ε, και να παρουσιάσουν έργο. Στο πλαίσιο του σημερινού πάνελ, εγώ θα σταθώ σε ορισμένα κενά και προκλήσεις που υπάρχουν. Κάποια έχουν ήδη αναφερθεί. Το πρώτο αφορά τη, τις διαδικασίες καθορισμού του καθεστώτος του ανεθαγενούς. Θα ήθελα εδώ να ε, υπογραμμίσω ότι σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ε, προσχωρήσει στην σύμβαση του 1954 για το καθεστώς των ανεθαγενών. Οι μοναδικές εξαιρέσεις εδώ είναι η Κύπρος, η Εστονία, η Μάλτα και η Πολωνία. Υπάρχουν αυτά τα κενά προσχώρηση. Αυτέ οι χώρε θα πρέπει να προσχωρήσουν. Θα ήταν ένα πολύ καλό επίτευγμα για την εκδήλωση που σα ανέφερα το 2019. Τα κράτη που έχουν προσφογράψει την Σύμβαση του 54 προφανώς έχουν υποχρεώσεις να δώσουν ένα, μια συγκεκριμένη αντιμετώπιση ε, στους ανθαγενείς. Ενώ δεν υπάρχει καμία ρητή υποχρέωση στη Σύμβαση του 54 για, για τη θέσπιση συγκεκριμένης διαδικασίας ε, για τους ανθαγενείς, ε, όμως αυτό υπονοείται προκειμένου να τους χορηγηθεί το νομικό καθεστώς το οποίο δικαιούνται. Γι' αυτό και μας προκαλεί έκπληξη και είναι σημαντικό κενό ε, στην εφαρμογή της νομοθεσίας, γιατί μέχρι σήμερα μόνο ε, ένας μικρός αριθμός κρατών μελών έχουν θεσπίσει τέτοιες ειδικέ διαδικασίες ε, προς διορισμού καθεστώτος ανθαγένειας. Οι χώρες που το έχουν κάνει είναι η Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Νομένα Βασίλειο, Ουγγαρία και Λετωνία αλλά πρέπει να γίνουν και άλλα για να ε, διασφαλίσουν ότι πρόκειται για αξιόπιστες, εύρωστες ε, διαδικασίες αυτές σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Σε ό,τι αφορά τους πόρους, κάποιος ανέφερε ήδη το εγχειρίδιο της υπερσαρμοστίας για τους ανεθαγενείς που ε, παρέχει συμβουλές για τον τρόπο διαμόρφωσης μιας ε, αξιόπιστης τέτοιας διαδικασίας και μάλιστα έχουμε προσθέσει και ένα νέο έγγραφο σε αυτό το θέμα, ε, ένα έγγραφο βέλτιστων πρακτικών για την ε, τον εντοπισμό των καλύτερων διαδικασιών αυτών. Ελπίζω αυτό να σας βοηθήσει καθώς θα προχωρείτε σε αυτή τη διαδικασία. Ένα από τα ζητήματα που δεν έχει συζητηθεί αρκετά, πιστεύω, σε ό,τι αφορά την χαμηλή κάλυψη των SDP στην Ένωση, είναι ότι οδηγεί αναγκάζει πολλούς να ε, ζητήσουν άσυλο ακόμα και αν δεν φοβούνται τη δίωξη. Όταν αυτό συμβαίνει ε, είναι αμοιβαία επιζήμια διαδικασία γιατί είναι και περί το άχθος ε, για τις αρμόδιες αρχές αλλά και για τους ανθαγενείς είναι, του ζημιώνει γιατί δεν έχουν τη νομική προστασία την οποία δικαιούνται και δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στις κοινωνίες τις οποίες διαμένουν. Μία σχετική πρόκληση είναι ε, το ευρύ φάσμα διαδικασιών που υπάρχει στο μεταναστευτικό πλαίσιο. Κάποιες χώρες καταγράφουν ορισμένα άτομα ως ανθαγενή με βάση το προσωπικό ισχυρισμό. Άλλοι βάση ε, τεκμηρίωσης της ανιθαγένειας που σπάνια βέβαια κατέχουν ε, η ίδια ανηθαγενείς και κάποια κράτη δεν έχουν καμία δυνατότητα να καταχωρήσουν κάποιον ως ανιθαγενή. Υπάρχει λοιπόν μια ε, ποικιλομορφία την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Μια ανησυχητικό εικόνα τώρα είναι ότι έχουμε δεκαπλάσιο αριθμό ατόμων που αιτούνται άσυλο και καταχωρίζονται ως αγνώστου ηθαγένειας. Στα 14 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, που χρησιμοποιούν ε, την κατηγορία αγνώστου ηθαγένειας, πήγαμε από τους 2.400 το 2012 σε πάνω από 20.000 ε, το 2016. Κάποια από αυτά τα άτομα σίγουρα είναι ενθαγενή για να τους δώσουμε την απαραίτητη προστασία που δικαιούνται, αλλά υπάρχει και ανάγκη για το κράτος να έχει ακριβείς πληροφορίες για το ποιος υπάρχει στην επικράτεια. Επομένως, η ικανότητα καταχώρησης των ατόμων ως ανιθαγενών θα πρέπει να υπάρχει σε όλη την Ένωση. Κάτι τελευταίο στο οποίο θα σταθώ ακροφηγώ είναι η έλλειψη ευαισθητοποίησης και κατανόησης για το καθεστώς των ανιθαγενών ε, μεταξύ του προσωπικού και των αρχών επιβολή του νόμου, αστυνομία, συνοριοφυλακή, ε, υπάλληλοι Frontex, νομική, διερμηνείς και ούτω καθεξής. Αυτό είναι ένα σημαντικό κενό το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσει το Κοινοβούλιο και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να προσθέσω εδώ Γι' αυτό το κενό είναι ότι οδηγεί σε παρανοήσει. Κάποιο ανέφερε τη λανθασμένη αντίληψη ότι η διαδικασία προσδιορισμού ε, του καθεστώτος ανεθαγένεια μπορεί να προσελκύσει άλλους μετανάστες. Τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτό δεν ισχύει. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση... Ε, μάλλον τα στοιχεία δείχνουν ότι το 2010 έχει μείνει σταθερό ο αριθμός, στα περίπου 200 άτομα κάθε χρόνο που ασκεί και επωφελείται αυτή τη ε, διαδικασία. Και σε άλλες χώρες που έχουν αυξημένο αριθμό μεταναστών και τούτον άσυλο, ο αριθμός των ανεθαγενών μένει μικρός και διαχειρίσιμος. Αυτά ήθελα να πω σε ό,τι αφορά την ε, ταυτοποίηση και την προστασία και τα κενά που υπάρχουν σε αυτού του τομεί. Δεν μίλησα ακόμα για την πρόληψη και τη μείωση δεν θα το κάνω, ε, απλώς ε, ήθελα να αναφέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει παροτρύνοντας όλα τα κράτη-μέλη να προσχωρήσουν και να ελοποιήσουν ε, καταλήλως τα πρότυπα της Σύμβασης του 1961 για την μείωση ε, των ανιθαγενών. Όπως ανέφεραν ορισμένοι, σήμερα εννέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν προσχωρήσει σε αυτή τη σύμβαση που έχει τα απαραίτητα εχέγγυα που αποτρέπουν την γένεια. Και προκαλεί έκπληξη το γεγονό, νομίζω το ανέφερε ενδεχομένω ο Κρί, ότι η υλοποίηση ακόμα και μεταξύ των ε, ε, συμβαλωμένων μερών των εχεγγύων αυτών δεν είναι η κατάλληλη και πιο ενδεδειγμένη. Υπάρχουν δύο βασικά στοιχεία. Πρώτον, όλοι να προσυπογράψουν και να προσχωρήσουν στη Σύμβαση του 61, αλλά εξίσου σημαντικό είναι όλοι να την υλοποιήσουν. Και αυτό δεν συμβαίνει σήμερα. Για παράδειγμα, ε, τα ηχέγγυα για όσου γεννιούνται στην επικράτεια και αλλιώ θα ήταν ανηθαγενεί να παίρνουν ηθαγένεια. Κάποια κράτη-μέλη ε, εφαρμόζουν αυτό το ηχέγγυο μόνο εάν οι γονεί ε, διαμένουν στη χώρα από την αρχή. Αυτό όμω δεν είναι η σωστή εφαρμογή τη σύμβαση. Κλείνω με τι εξή τέσσερι συστάσει. Πρώτον, τα κράτη-μέλη που, που δεν έχουν προσυπογράψει τη σύμβαση ανηθαγένεια θα πρέπει να τα παροτρύνουμε για να προσχωρήσουν. Σύμφωνα και με τη δέσμευση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην ε, υψηλού επίπεδου συνάντηση του 2012 στη Νέα Υόρκη, από τότε δεν, καμία άλλη χώρα δεν προσυπέγραψε την σύμβαση του 1954 και αυτό είναι απογοητευτικό. Δεύτερον, όλα τα κράτη-μέλη που δεν έχουν κατάλληλε και ξεχωριστέ διαδικασίε διορισμού του καθεστώτο ανεθαγένεια θα πρέπει να ε, τι υιοθετήσουν και εμεί είμαστε στη διάθεσή για να σα στηρίξουμε σε αυτή τη διαδικασία. Τρίτον, τα κράτη μέσα Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κληθούν να ενισχύσουν ε, τη διαδικασία ταυτοποίηση των ανθαγενών ε, στο πλαίσιο των υφιστάμενων συστημάτων καταχώρησης. Θα πρέπει να επιτρέπουν λοιπόν την καταγραφή κάποιου ως βάσει του ισχυρισμού του ίδιου του προσώπου, όπως ισχύει και για την ηθαγένεια. Και οι πάλι το προσωπικό θα πρέπει να λάβουν γνώση της ανηθαγένειας και τέτοια κατάρτιση θα πρέπει να παρέχεται διαδεδομένα ε, στο πλαίσιο άλλων καταρτήσεων για το άσυλο, τις επιστροφές ε, και την προστασία των δεδομένων και των δικαιωμάτων. Τέταρτον, Όλοι, όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν σημαντικό ρόλο να δραματίσουν για να παροτρύνουν, να ενθαρρύνουν ε, ε, την ε, λήψη σημαντικών μέτρων και θετικών μέτρων εν ώψη τη συνάντηση του 2019. Ισχυρέ διπλωματικέ σχέσει και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών θα είναι εξαιρετικά σημαντικέ για την επιτυχή ε, διοργάνωση αυτή τη εκδήλωση και γενικά τη εκστρατεία τη ΥΠΑ Αρμοστία για του πρόσφυγε συνολικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ συγκεκριμένε οι παρατηρήσει σα και χρήσιμε μας μόνο τώρα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Και πάλι αν μπορείτε να μείνετε στα 6-7 λεπτά, βλέπετε ότι έχουν αποχωρήσει περισσότεροι συνάδελφοι. Αν μπορείτε να μείνετε στα 6 λεπτά, καλύτερα. Αλλιώς θα μιλάτε μόνο σε μένα, που εγώ δεν έχω πρόβλημα. Βέβαια υπάρχει και μετάδοση μέσω διαδικτύου. Καλό είναι όμως να υπάρξουν κάποιες, να κάποιες ερωτήσεις στο τέλος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο. Αξιότιμοι βουλευτέ, κυρίε και κύριοι, συνάδελφοι, θα προσπαθήσω σε έξι λεπτά να προσπαθήσω να σα τα πω αυτά που είχα προγραμματίσει να σα τα πω σε δέκα λεπτά. Για να δούμε. Οπότε α επικεντρωθούμε στα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στου ε, ανιθαγενείς. Δηλαδή για να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτή η προστασία. Κάνουμε επομένω ε, να δούμε αυτή την ε, παρουσίαση από πλευρά νομική. Είναι κάπω τεχνικό το θέμα, συμπαράτε με. Τέλο πάντων, για να δούμε ποια είναι η νομική φύση του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων τη Ένωση. Από την συνθήκη τη ε, Λισαβόνα τέθηκε σε ισχύ, είναι πρωτογενέ δίκαιο και έχει άμεση ισχύ και κάθετη ισχύ σύμφωνα με το δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ήδη έχει δημορφωθεί νομολογία ΑΠ, δεν δουλεύει το τηλεχειριστήριο. Ανάτο, εντάξει. Μπορεί να παρακολουθήσω αυτά που λέω, είναι πιο εύκολο με τις διαφάνειες. Πρωτογενές, δευτερογενές δίκαιο και οι διεθνείς συνθήκες θα πρέπει να συνάδουν με όλα αυτά. Αυτό είναι το νομοθετικό πλαίσιο και βέβαια και η ερμηνεία του σε αυτό το νομικό πλαίσιο και του. Επόμενη διαφάνεια. Για να δούμε τώρα με δύο λόγια τι γίνεται με την εμβέλεια του χάρτη. Όπως βλέπετε, δεσμεύει τα θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή του κοινωτικού δικαίου. Βέβαια, η νομολογία του ΔΕΚ προστίθεται σε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Όσον αφορά τώρα την ερμηνεία του χάρτη, θα πρέπει αυτό να γίνεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έτσι θα πρέπει να δίνεται η ερμηνεία και σύμφωνα με την ομολογία του Δικαστηρίου ή της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Στρασβούργου. Επίσης, ακόμη ένα επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων είναι ότι κανένα δικαίωμα του χάρτη θα πρέπει να ερμηνευθεί ως περιοριστικό άλλων δικαιωμάτων, άλλων συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πάμε δύο διαφανείς πιο κάτω και βλέπουμε τώρα σε σχέση με τους ανιθαγενείς τι προβλέπει το ευρωπαϊκό δίκαιο. Μόνο άμεσα ρυθμίζεται το φαινόμενο και σποραδικά. Αλλά το ίδιο ισχύει και στην σύμβαση της Νέας Υόρκης του 54. Αυτό είναι α, δευτερογενές ευρωπαϊκό δίκαιο. Να δούμε κάποια παραδείγματα. Τι γίνεται με την προστασία τους. Έχουμε τον συντονισμό των ε, προγραμμάτων και πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης. Επίσης, αναγνωρίζεται η κίνηση προσώπων, διακίνηση προσώπων χωρίς θεώρηση διαβατήρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε επίσης σχετική νομολογία του ΔΕΚ για την προστασία των ανιβαγενών. Όχι επομένως περιστολή των αριθμών τους, αλλά προστασία. Έχουμε τη σχετική απόφαση εδώ, όσον αφορά το ότι δικαιούνται Παλαιστίνοι, που ζούσαν στον Λίβανο λέει ότι μπορούν αυτοί που είχαν πάει στην Γερμανία τότε να έχουν κάποιες απολαβές κοινωνικής πολιτικής, κάποια κοινωνικά επιδόματα. Με την συνθήκη της Λισαβόνας προέκυψε και κάτι άλλο όπως είπαν και οι ομιλητές. Υπάρχει σχετικό άρθρο στη Συνθήκη Λειτουργία Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέει ότι θα πρέπει να θεωρούνται υπήκοοι τρίτων χωρών όσον αφορά τους συνολικούς ελέγχους και τα σύναφη. Τώρα παρακάτω, για να δούμε πώς ο χάρτης μπορεί να παράσχει συγκεκριμένη προστασία. Τώρα, η εμβέλεια του πεδίο εφαρμογής ε, περιέχει διάφορα δικαιώματα του χάρτη και λέει ότι ανεξαρτήτως ηθαγενείας αυτά τα δικαιώματα ισχύουν για όλους. Ε, Αξιοπρέπεια, δικαίωμα στη ζωή, στην σωματική ακαιρεότητα, ελευθερία και ευγενική ζωή, μη διακρίσεις, ε, το δικαίωμα προσφυγής στα δικαστήρια και σε ένδικα μέσα. Επομένως, βλέπετε τώρα αυτήν την απαρίθμηση των δικαιωμάτων που σας ανέφερα προηγουμένως εντάχει. Και σας τονίζω δύο εξ αυτών που ενδιαφέρουν τώρα. Η, το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια σε σχέση με την κράτηση, περισμό της ελευθερίας δηλαδή των ανιθαγενών. Το επόμενο, επόμενη διαφάνεια παρακαλώ, το ε, δικαίωμα αποφυγής δυσμενών διακρίσεων. Από τον Δεκέμβριο του 2015 Ανεγνώρισε το Συμβούλιο ότι θα πρέπει να προστατευτούν τα δικαιώματα των προσώπων αυτών και να περισταλεί ο κίνδυνος των δεσμενών διακρίσεων και αναγνωρίζει την ισότητα μεταχείρισης. Εδώ πρώτα-πρώτα έχουμε έναν κατάλογο δυσμενών διακρίσεων και των αιτιών τους. Βέβαια δεν είναι αποκλειστική η σχετική επαρρύθμιση και αφορά πάσα δεσμενή διάκριση, αλλά κάποιο μπορεί να πει ότι αυτό ισχύει για την σχέση μεταξύ ανιθαγενών και λοιπόν προσώπων, είτε υπηκών ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε τρίτων χωρών. Η άλλη, η επομένη παράγραφος, λέει για τα της ηθαγένειας. Ρητός το προβλέπει, αλλά δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτού του είδου δηλαδή διάκριση από τη βάση τη ηθαγένεια. Για του υπηκόου τρίτων χωρών και του ανηθαγενεί. Επομένω εδώ έχουμε μια πιθανή, μια λιθοφανή, τέλο αξιοπρεπή ερμηνεία, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί από το δικαστήριο. Επίσης, έχουμε την ερμηνεία του Δικαστήριου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όσον αφορά την εθνικότητα και την σχετική δυσμενή διάκριση. Άρα και εδώ έχουμε κάτι που μπορεί να μας βοηθήσει. Επίσης, είχαμε αυτή την πρωτοβουλία των πολιτών όσον αφορά το Minority Safe Pack για την προστασία των μειονοτήτων στην Ένωση και οι συντάκτες αυτής της πρωτοβουλίας επίσης πρότειναν την τροποποίηση της δευτερογενούς νομοθεσίας και του κοινοτικού δικαίου, τόσο ώστε να καλύψει και τους ανηθαγενείς. Τέλος πάντων, τώρα είναι στη φάση της συλλογής υπογραφών, αλλά θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δει τι θα κάνει σχετικά με αυτό. Τώρα, πριν ολοκληρώσω, να σας πω το εξής με αυτή την διαφάνεια πόσο ο χάρτης μπορεί να προστατεύσει τους ανηθαγενείς από αυθαίρετη παράνομη κράτηση. Είπα, είπαμε τα υπόλοιπα και πάμε κατευθείαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιστροφή, επαναπατρισμό ενδεχομένω. Είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει η εύλογη πιθανότητα, μάλλον θα πρέπει να σταματήσει η κράτηση όταν δεν υπάρχει κάποια εύλογη πιθανότητα απομάκρυνσης. Αυτό είναι κλασική περίπτωση για του ανεθαγενεί. Πάντω τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να πάυσουν την κράτηση. Εάν ισχύει αυτό που προαναφέραμε. Επίσης, το ΔΕΚ στην ομολογία αναφέρεται στο ότι θα πρέπει εν στενή ενία να νοείται η κράτηση και στέλνηση ελευθερίας ενός προσώπου. Δεν έχουμε χρόνο για το με την επόμενη διαφάνεια και πάμε στην τελευταία. Θα πρέπει να δούμε πώς η υπηρεσία με τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει βοηθήσει μέχρι τώρα. Υπάρχουν κάποιες ε, έμεσες ε, ενέργειες που έχουν γίνει για τους ε, και όπως είδαμε και στα άλλα παραδείγματα έχουμε αυτές τις διαδικασίες, τη σχετική έκθεση για τους ανηθαγενείς. Πριν από 7 χρόνια, πριν από 3 χρόνια είχαμε αυτό το εγχειρίδιο και υπάρχει ένα σχετικό ε, χωρίο εκεί, ένας ε, από παράγραφο εδάφιο και λέει ότι θα πρέπει ήταν για κάποιους κουβετιανούς στα ελληνικά νησιά και έλεγε το πώς θα πρέπει να ενημερώνονται αυτές οι ομάδες στα hot spots, στα κέντρα υποδοχής. Δεν θα πρέπει να υπάρχει de jure και de facto αυθαίρετη ε, κράτης και στέρες ελευθερίας αυτών και επίσης είπαμε ότι θα πρέπει αυτό το θέμα να ενσωματωθεί στην αξιολόγηση των αποστολών Σέγγεν. Και να ερμηνεύσουμε αυτή την νομική έννοια, την έλλειψη εύλογης ε, πιθανότητας ε, με απομάκρυνσης. Ξέρω ότι υπερεύουν τα όρια που θέσατε, Πρόεδρε, αλλά τέλο πάντων είμαι έτοιμο να απαντήσω τυχόν ερωτήσεις. Μας μένει ένα ακόμη ομιλητή πριν να μπορέσουν να κάνουν παρατηρήσει ή ερωτήσεις τα μέλη μας. Ο κύριος Νάσ και πάλι, ο οποίο θα μιλήσει για αυθαίρετη κράτηση. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Δεν είναι τεχνική η παρουσίασή μου. Να σας πω λίγα για τον εαυτό μου πρώτα. Άρχισα να δουλεύω για θέματα ανιθαγένειας το 2010 σε μια μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο με στόχο να βάλει το Ηνωμένο Βασίλειο σχετική νομοθεσία. Από το 2011 που παντρευθήκαμε με τη γυναίκα μου έχουμε ε, περάσει διάφορα. Το 2010 ο γιος μου γεννήθηκε την ίδια ημέρα, στις 25η ε, επέτειο το, της διακήρυξης δικαιωμάτων των παιδιών. Μετά άρχισα να ασχολούμαι με άλλα θέματα. Ε, ξεκινήσαμε το ENS μαζί με την Λόρα. Έχω επισκεφθεί ε, καταπληκτικούς τόπους από το 2010 και έχω συναντηθεί με πάρα πολύ εντυπωσιακούς ανθρώπους έχω ε, περάσει διάφορα. Πάντως, εν τέλει η ψήφος μου που ήταν υπέρ του να παραμείνει η χώρα μου στην Ένωση δεν μπόρεσε να μεταστρέψει. Όλα αυτά τα χρόνια, ε, τα 7 τελευταία χρόνια, είδατε πόσα πράγματα πέρασα. Ε, τα 7 χρόνια είναι πολλά χρόνια στη ζωή ενός ανθρώπου. Για φανταστείτε λοιπόν να προσπαθήσετε τώρα να σβήσετε τα 7 χρόνια από τη μνήμη σας, να τα αντικαταστήσετε με μια καθημερινότητα χωρίς καμία αλλαγή, με απογοήτευση, με απελπισία, με ε, ψυχολογικά τραύματα, όλα τα πράγματα που δεν θα μπορούσατε να κάνετε και σκεφτείτε τον Άντων ο οποίος ε, πέρασε από κράτηση 7 χρόνια στη Βουλγαρία διότι δεν του προσφέρθηκε καμιά προστασία ως αν θα κρίση, σε παρακαλώ, είναι λίγο πιο αργά. Δεν θα σε διακόψω, αλλά καλά θα είναι να σε προλαβαίνουν οι διερμηνείς. Οι διερμηνείς ε, ευχαριστούν τον Πρόεδρο για την παρατήρησή του. Τα 7 χρόνια λοιπόν είναι πολύ καιρό και για μερικού μάλιστα είναι και περισσότερα από 7 χρόνια. Ιστορίε όπω του Άντων συμβαίνουν σε πολλέ χώρε, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και ο Άντων είναι ένα από τα πρόσωπα στα οποία μιλήσαμε για την έκθεσή μα προστασία ανιθαγενών από την αυθαίρετη κράτηση. Στα λίγα λεπτά που μου μένουν θέλω να μιλήσω για τους λόγους για τους οποίους οι ανιθαγενείς κινδυνεύουν να κρατηθούν αυθαίρετα. Και τι μπορεί να γίνει για να αντιμετωπιστεί αυτός ο κίνδυνος. Δείξτε μου την επόμενη διαφάνεια. Έχω ένα παράθεμα από τον Φρανσουά Κρεπό, ειδικό ε, εισηγητή για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών. Είπε λοιπόν ότι η κράτηση των μεταναστών είναι μία από τις ε, σιωπηρές τραγωδίες που πλήττουν τους ανθρώπους πίσω από κλειστές πόρτες, μακριά από τα βλέμματα των δημοσιογράφων, αλλά με το ανθρώπινο κόστος. Και συνεχίζει λέγοντας ότι πρόκειται για μια τραγωδία η οποία είναι δυνατόν να αποφευθεί, αλλά λόγω της έλλειψης πολιτικής θέλησης πλήττει χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο. Επόμενη διαφάνεια. Για το λόγο αυτό το 2015 η οργάνωσή μου άρχισε ένα πρόγραμμα τριετίας για να ε, βοηθήσει να αντιμετωπιστούν οι αυθαίρετες κρατήσεις ε, ανιθαγενών. Σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη έχουμε δημοσιεύσει εκθέσεις για έξι χώρες, τις οποίες βλέπετε στην οθόνη, με μεθοδολογία η οποία περιλαμβάνει και έρευνα αλλά και ε, συνεντεύξεις με τους ίδιους τους κρατουμένους. Τον προηγούμενο μήνα προχωρήσαμε ένα βήμα παραπέρα. Κάναμε μια, συνέντε, μια συνάντηση στην Βουδαπέστη με 120 συμμετέχοντε από 30 ευρωπαϊκέ χώρε και ξεκινήσαμε αυτό που λέμε Agenda for Change και, ε, μια ολόκληρη εκστρατεία. Το κοινοβούλιο εκπροσώπησε η Jean Lambert, Ευρωβουλευτή, η οποία τόνισε μερικού από του τρόπου που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το πρόβλημα αυτό και θα επανέλθω σε λίγο την επόμενη διαφάνεια. Η κατάσταση την οποία περιγράφει ο Φαρίντ στην διαφάνεια που βλέπετε θα είναι γνωστή και σε άλλους. Οι εμπειρίες ανδρών και γυναικών με τους οποίους μιλήσαμε δείχνει την έλλειψη εμπιστοσύνης στα νομικά συστήματα. Υπάρχουν κάποιες καλές πρακτικές, αλλά συνήθως δεν εφαρμόζονται. Η αυξανόμενη χρήση της αυθαίρετης κράτησης σε βάρος μεταναστών είναι μια τάση παγκόσμια και ευρωπαϊκή και κυρίως πλήττει ανιθαγενείς, οι οποίοι δεν έχουν χώρα στην οποία να μπορούν να επιστραφούν και οι άνθρωποι αυτοί περνούν από επανειλημμένες αυθαίρετες κρατήσεις. Βασικό συμπέρασμα της έκθεσής μας Agenda for Change είναι η παράληψη των χωρών να εντοπίσουν τους ανιθαγενείς και επομένως να τους προσφέρουν την κατάλληλη προστασία στην ουσία η πρακτική της ε, ε, κράτησης σε βάρος μεταναστών οφείλεται στην έλλειψη εντοπισμού του στοιχείου της ανιθαγένειας. Όπως τα είπε σωστά η Μέλανη πριν από λίγο, η μεγάλη πλειοψηφία των χωρών μελών δεν έχουν συγκεκριμένες διαδικασίες για τον καθορισμό της ανιθαγένειας ή τρόπο για να ε, διορθωθεί αυτό. Το αποτέλεσμα αυτών των συστημικών παραλήψεων είναι οι ανιθαγενείς να παραμένουν χωρίς νομικό καθεστώς, χωρίς να έχουν το δικαίωμα να εργαστούν, εκτός κοινωνικής προστασίας. Οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζουν απομόνωση, μεγάλο κίνδυνο εκμετάλλευσης και εγκληματικότητας επιβίωσης. Για να, πρέπει να σπάσει αυτός ο φαύλος κύκλος και για να γίνει αυτό χρειάζεται επίγουσες αλλαγές στην νομοθεσία. Η δική μας Agenda for, for Change και στην έκθεσή της προ, προτείνουμε πέντε συστάσεις για το πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό ώστε να προσφερθεί καλύτερη προστασία σε ανθρώπους, στους ανθρώπους, σε ανηθαγενή πρόσωπα δηλαδή. Πρώτον, χρειάζεται να υπάρχουν εναλλακτικέ επιλογές στην κράτηση. Για παράδειγμα, Βουλγαρία και Μάλτα προχωρούν αυτόματα σε κράτηση ενός ατόμου όταν δεν είναι δυνατόν να επιστραφεί. Αυτό εξηγεί πως ο Άντων, τον οποίο ανέφερα προηγουμένως, κατέληξε να περάσει 7 χρόνια σε κράτηση. Και η παράληψη αυτή είναι κοινή σε όλη την Ευρώπη και παρά το γεγονός ότι εναλλακτικέ επιλογές δεν είναι περισσότερο δαπανηρές, είναι όμως περισσότερο ανθρώπινες. Δεύτερο, όλες οι χώρες θα χρειαστεί να προβλέψουν συγκεκριμένες διαδικασίες για τον καθορισμό του καθεστώτος του κάθε προσώπου. Τα είπα αυτά η Μέλανη προηγουμένως. Χωρίς διαδικασίες αυτές, οι χώρες που δεν είναι σε θέση να εντοπίσουν ποιος ε, που διαβεί στην επικράτειά τους πρέπει να χαίρει τις προστασίες της ε, ε, σύμβασης του 1954, δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2015 δίνουν ξεκάθαρες κατευθύνσεις στις χώρες μέλη για να βελτιώσουν τις πρακτικές αναγνώρισης και ιδίως σε ό,τι αφορά την υποστήριξη από την πλατφόρμα ανιθαγένειας του EMN. Παρόλο όμως που υπάρχουν χώρες μέλη που δεν έχουν τέτοιες διαδικασίες, οι αξιωματούχοι της μετανάστευσης καλούνται να εντοπίσουν τα πρόσωπα που κινδυνεύουν από αυτό. Τρίτη σύσταση, για να μην είναι η κράτηση αυθαίρετη θα πρέπει να μην αποτελεί δυσμενή διάκριση. Και αυτό θα πρέπει να ισχύει για όλες τις χώρες. Σε πολλές όμως χώρες δεν συμβαίνει αυτό. Τέταρτη σύσταση είναι κρίσιμο να διευκολυνθεί η ένταξη στην κοινότητα, ιδίως προσφέροντας τρόπους, προσφέροντας οδούς για την τακτοποίηση των ε, προσώπων, ε, πρόσωπα τα οποία συχνά χωρίς να φταίνε δεν μπορούν να συμβάλλουν στη ζωή της κοινότητας. Έχουμε πολλές ιστορίες ανδρών και γυναικών που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο αυτό. Ιδίως με απασχόλησε η περίπτωση του Κριστόφ, ενός ανιθαγενού στην Βουλγαρία, που μου λέει «Είμαι εδώ 24 χρόνια, όχι μήνες ή ώρες, 24 χρόνια». Και η κράτηση ήταν η πιο βαριά και ταπεινωτική τιμωρία που υπέστη στη ζωή μου. Πέμπτο, χρειάζεται καταγραφή, διότι η έλλειψη ε, συγκεκριμένων δεδομένων δεν επιτρέπει και οι να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Η ανηθαγένεια πρέπει να καταγράφεται με ακρίβεια και να αναλύεται. Ορισμένες από τις παραπάνω δράσεις πρέπει να αναλυθούν από εθνικές αρχές. Υπάρχει όμω καθαρό ρόλο και για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για παράδειγμα, πρόσφατε τροπολογίε που προτάθηκαν για τον κανονισμό διαδικασιών ασύλου προβλέπουν τα σχετικά. Το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να ζητήσει επίσης τον κανονισμό των Migration Statistics να τροποποιηθεί για να επιβάλλει στις χώρες μέλη να καταγράφουν τους αριθμούς ανιθαγενών που διαβιούν στις επικράτειές τους. Και για να βελτιωθεί η παρακολουθήση, το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει ανα διετία, ε, υποβάλει έκθεση για την πρόοδο που ε, γίνεται στην ε, συγκεκριμένη ε, διαδικασία. Το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης το οποίο αναφέρθηκε ο Κλόντ προηγουμένως θα μπορούσε να προβλέψει και μια ειδική λύση για την ανιθαγένεια. Επόμενη διαφάνεια. Θέλω να οκλώσω την παρουσίασή μου με την ιστορία του Ρόμαν που την έχουμε περιλάβει στην έκθεσή μας Still Stateless, Still Suffering το 2014. Ο Ρόμαν ανιθαγενής δεν μπορούσε να κληρονομήσει την ε, ε, ηθαγένεια ούτε από τον πατέρα του πρώην Ιουγκοσλάβου ούτε από τη μετέρα του πρώην κάτοικο της Σοβιετικής Ένωσης. Κατέληξε στην Σλοβακία στις αρχές της δεκαετίας του 90. Δεν είχε όμως ούτε το καθεστώς του πρόσφυγα, ούτε άλλη μορφή προστασίας. Και επειδή η Σλοβακία δεν έχει ε, μηχανισμό προστασίας για τους ανηθαγενεί παρέμεινε παράνομα στη χώρα και διαβιούσε στους δρόμους. Οι αρχέ ποτέ δεν μπόρεσαν να τον απελάσουν παρόλο που το αποπειράθηκαν πολλές φορές. Συνελήφθη πάνω από 25 φορές και πέρυσε πολλούς μήνε σε κράτηση. Τα τελευταία 20 χρόνια δεν μπόρεσε καν να παντρευτεί διότι δεν ρυθμίστηκε ποτέ η περίπτωσή του. Δυστυχώς το 2015 απεδίωσε ο Ρόμαν μόνος του και σε απελπισία και ούτε καν δέχθηκαν να του ε, κάνουν μια αξιοπρεπή κηδεία. Η ιστορία του ε, Ρόμαν δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα και άλλα άτομα όμως που υπάρχουν δεν πρέπει να καταδικαστούν σε τέτοιου είδους διαβίωση. Το γεγονός ότι διαξάγεται σήμερα η παρούσα ακρόαση δίνει ένα σήμα ελπίδας. Ευχαριστούμε πολύ. Εξαιρετική αυτή η παρέμβαση. Πριν δώσουμε το λόγο στα τρία μέλη της Επιτροπής, ε, τους οποίους και ευχαριστώ, λέω ξανά και ξανά ότι είναι πέμπτη απόγευμα. Ήθελα μόνο να πω και η κυρία Βίξτρον θα ήθελε να το αναφέρει, γιατί είστε όλοι ειδικοί στο θέμα της ανηθαγένειας και κατανοείτε το πεδίο αυτό και τη διασύνδεσή του με πολλούς άλλους τομείς Είναι αφρηγουμένου κάτι τέτοιο στην Επιτροπή μας. Ο αριθμός των ακροάσεων που διοργανώνουμε, των προτάσεων σε μη νομοθετικό πλαίσιο, είναι πραγματικά ανεφρεγουμένου. Αντί λοιπόν να δούμε κατά πόσο θα υπάρχει μεγάλη ε, προσέλευση και τα λοιπά, ποια μέρα θα είναι. Είναι σημαντικό να διοργανώνονται παρόλα αυτά, γιατί σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει και συνέχεια, παρακολούθηση και από το δικό μας θεσμικό όργανο. Και εγώ στηρίζω μία ΜΚΟ που εργάζεται σε αυτό το τομέα της ανηθαγένειας ανηλίκων. Ευχαριστώ τον ε, Κρίς για όλη τη δουλειά που κάνει και το Ευρωπαϊκό ε, Δίκτυο Μεταναστών, αλλά και όλους τους ομιλητές που πήραν το λόγο σήμερα για τις εξαιρετικές τους παρεμβάσεις. Και συγγνώμη που σας πίεσα με τον χρόνο, αλλά έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να καταλήξουμε σε καλά συμπεράσματα, το οποίο θα μεταφέρω στους συντονιστές. Άντρη, θες να σχολιάσεις πρώτος και μετά να δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους. Ευχαριστώ. προς τον Κρίσνας να τον ευχαριστήσω για την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία. Ακόμα μία πρωτοβουλία εκρεμεί στην Επιτροπή Αναφορών για την Ανεθαγένεια με πάνω από 20.000 ε, άτομα που την υπέγραψαν πέρσι από τη Λετωνία και την Εστονία για να λυθεί το ζήτημα των μη πολιτών ε, της Εστονίας και της Λετωνίας και να τους χορηγηθούν δικαιώματα. Θεωρείτε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να στηρίξει αυτή την ε, πρωτοβουλία. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Πολύ σαφές ε, και συγκεκριμένο ερώτημα. Ε, κυρία Στάνοφκα, θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Δεν χρειάζεται βέβαια. Εντάξει, όχι τόσο να ρωτήσω. Να κάνω μια πρόταση θέλω για την αξιολόγηση της σημερινή ακρόασης. Βεβαίως να ευχαριστήσουμε όλους ε, τους ομιλητές και του δεύτερου πάνελ και ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε τον κύριο Κρίς Νάς και εγώ ήμουν εισηγήτρια για τον Οργανισμό Θεμελιωτών Δικαιωμάτων. Εκτιμώ τα όσα μας αναφέρατε, αλλά ακόμα παραμένει αυτό το πρόβλημα του άρθρου 51 στην εφαρμογή της χάρτας. Και θα ξέρετε κι εσείς ότι αυτό περιορίζει σημαντικά τις δυνατότητες που μας παρέχει η χάρτα, ιδίως στην Επιτροπή Αναφορών, που πρέπει να παραπέμψουμε στη χάρτα. Μετά έρχεται η Επιτροπή και μας λέει «Εντάξει, αλλά δεν είναι δική μας αρμοδιότητα». Είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χάρη εξαιτία μάλλον του άρθρου 51. Μια πολύ καλή έκθεση για την περαιτέρω εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Ε, εξαιτία του Brexit, η έκθεση δηλαδή Verhofstadt, μία από τις προτάσεις είναι να ε, καταργηθεί το άρθρο 51. Ιδίω επειδή ένα από τους ε, συντάκτε αυτού του άρθρου ήταν Βρετανό. Αυτό είναι το πρόβλημα λοιπόν. Γι' αυτό προτείνω στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, εφόσον πρόκειται για μια κοινή ακρόαση, να πάει ακόμα πιο πέρα και να συντάξει μια έκθεση δύο πρωτοβουλία ή να στηρίξει αυτή την αναφορά ε, για να περάσει είναι μια πρωτοβουλία που γίνεται κάθε χρόνο. Έτσι κι αλλιώς πολύ λίγα προβλήματα αντιμετωπίζουμε. Το θέμα της διάσχεσης διέλευσης των συνόρων και μερικά άλλα. Δεν καλύπτεται όμως η ενθαγένεια. Ας συζητήσουμε εκ νέου το θέμα της ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Έχει έρθει η ώρα. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να λύσουμε αυτό το θέμα της ανηθαγένειας, ιδίως των ανηλίκων, αξιοποιώντας ε, την ε, ε, πρακτική εφαρμογή της έννοιας της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Γιατί όχι. Να αξιοποιήσουμε και τους εξαιρετικούς συμπληρογνώμενους που έχουμε εδώ σήμερα, να αναζητήσουμε μία πρόταση για να υλοποιήσουμε αυτό το όραμα της Ευρωπαϊκής Σε Ευχαριστούμε. Κυρία Βαρζία δεν θέλει να πάρει το λόγο. Την ευχαριστώ όμως ε, που έμεινε μέχρι το τέλος της ακρόασης. Είναι σημαντικό Δεν ξέρω αν θέλουν οι ομιλητές να πάρουν το λόγο, γιατί ε, συμπερασματικά εγώ θα αναφέρω κάποιες μελλοντικέ κινήσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πολλά ερωτήματα απευθυνθήκαν προς εμένα, οπότε θα ήθελα να απαντήσω. Στο πρώτο ερώτημα μπορώ να πω ότι η δική μου γνώμη μάλλον δεν έχει μεγάλη σημασία. Ερωτήσατε κατά πόσο πρέπει να στηρίξουμε αυτή την... Ε, αν υπάρχει, πρέπει να υπάρχει μια αναφορά για τα θέματα της κράτησης, σαφώς. Και η σημερινή ακρόαση αναδεικνύει την ε, σημασία των αναφορών, ε, γιατί και αυτό το θέμα ξεκίνησε από μια αναφορά. Είναι σημαντικό λοιπόν για τέτοια θέματα όπως είναι η Θαγένεια. Μετά, και με βάση την εξαιρετική κάτια που, απάντησε που έδωσε προηγουμένω έχουμε αυτή την κατάσταση. Είτε δηλαδή κάποιοι είναι υπήκοοι, είτε ανηθαγενείς. Είναι μυθοπλασία κάποιος από νομική άποψης να ισχυρίζεται κάτι διαφορετικό και είναι πολύ επικίνδυνο και από πλευρά Ευρώπης ε, να ισχυριζόμαστε κάτι τέτοιο γιατί μπορεί να δίνει ιδέε σε άλλες ε, χώρε που θέλουν να διαγράψουν ένα τμήμα του πληθυσμού του για διάφορους λόγους. Αυτό δεν σημαίνει όμως ε, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να προχωρήσει το θέμα της ε, αναθέμα ξεχωριστά δηλαδή. Ακούσαμε ε, πολλές λύσεις και προτάσεις, μπορεί να τις συνοψίσει και ο Πρόεδρος. Εμείς θα θεωρούσαμε χρήσιμο όχι μόνο να έχουμε μια ε, ειδική στρατηγική, αλλά και ένα ειδικό ψήφισμα για αυτό το θέμα που θα εντοπίζει τυχόν άγουσες ανάληψης δράσης και θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε αυτή την ολιστική προσέγγιση που δεν έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Στανόφκα, νομίζω ότι τα περισσότερα σχόλια ε, και μια έκκληση προς την ε, ΛΥΜΠΕ να εργαστεί πιο σκληρά για την Ευρωπαϊκή Εθνογένεια μας τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ τον Κρίς και βέβαια όλοι οι ομιλητές ήταν εξαιρετικοί. Η Επιτροπή Αναφορών αρχικά. Είπατε ότι η Επιτροπή Αναφορών είναι αξιόλογη γιατί αποδεικνύει την αξία της ξανά και ξανά είναι πολύ σημαντική επιτροπή για τέτοιου είδου πολύπλοκα ζητήματα και οδηγούν στη οργάνωση τέτοιων ε, δημοσίων ακροάσεων. Και θέλω να τους ευχαρώ που κάνουν όλη τη δουλειά σε ένα πολύ ε, δύσκολο περιβάλλον. Κάποια ανέφεραν για τα ζητήματα της Αγένεια εν μέσω Brexit. Αυτό είναι ένα παράδειγμα μόνο. Δεν είμαι ειδικό στα ζητήματα της Επιτροπής ε, Αναφορών, αλλά έχουμε πολλά κοινά μέλη τη ΛΥΜΠΕ και τη ΠΕΤΗ. Ευχαριστώ λοιπόν την ε, Σεσίλια και του συναδέλφου από την Επιτροπή Αναφορών. Πρέπει να αξιοποιήσουμε το εργαλείο της Επιτροπής Αναφορών ε, όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, αυτό που σκεφτόμουν εγώ είναι ότι είναι ένα εξαιρετικά τεχνικό, ε, νομικίστικο ζήτημα, βέβαια και με μια σημαντική ανθρώπινη διάσταση, όπως πολύ σωστά ε, ανέφεραν οι μολυτές. Και μετά η διασύνδεση με άλλους ε, τομείς δικαίου, όπως το άσυλο και το καθεξής, περιπλέκει τα πράγματα. Όμως αυτή η πολυπλοκότητα δεν θα πρέπει να μας εμποδίζει πρέπει να καταλήξουμε σε μια στρατηγική, να υιοθετήσουμε ένα ψήφισμα, όπω είπε και ο Κρίς. Και να λάβουν υπόψη τα όσα κάνουν διάφοροι οργανισμοί, η Πατιαρμοστία για του πρόσφυγε, τα διάφορα δίκτυα, αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτά που πρότεινε η UNICEF. Γι' αυτό και εμεί ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια, γιατί θέλαμε να δούμε τι ρόλο μπορεί να αναλάβει το Κοινοβούλιο με τον ρόλο του ως ε, συνομοθέτη. Προτείνω λοιπόν στους συντονιστές μας να μαζί με την κυρία Βίκστρομ που είναι επίσης ιδιαίτερα έμπειρο μέλος ε, της ε, ΛΥΜΠΕ, να παρουσιάσουμε λοιπόν μια στρατηγική για να ε, προσδιορίσουμε την ανηθαγένεια ως ξεχωριστό σημείο. Δεν δεσμεύομαι βέβαια σε τίποτα, δεν υπόσχομαι τίποτα. γιατί η γραμματεία μου κοιτάζει λίγο στραβά. Επομένω, πολύ προσεκτικά μπορώ να αναφέρω ότι θα υπάρξει, θα δοθεί συνέχεια, αλλά με μια ολιστική προσέγγιση προς την ε, μετανάστευση. Προσπαθούμε ακόμα να τα εξετάσουμε από κοινού. Δεν έχει νόημα να σπάσουμε το θέμα της μετανάστευσης σε ξεχωριστά κομμάτια. Υπάρχει βέβαια και το θέμα της υλοποίησης που είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, από εδώ και πέρα έχουμε σημειώσει όλες τις απόψεις και η ε, συνεδρίαση αυτή, ε, καθώς και οι παρεμβάσεις των ομιλητών και των μελών έχουν διαδοθεί και μέσω διαδικτύου. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε πώς το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ μπορούν να σημειώσουν πρόοδο σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα ε, διατηρώντας βέβαια την επαφή και συνεργασία με την Επιτροπή Αναφορών. Και θα το δώσουμε όλα αυτά στους συναδέλφους. Όμως θέλω πρώτα να το συζητήσουμε με τους συντονιστές. Και με τα έμπειρα μέλη της Επιτροπής μας. Δεν θέλω να πω άλλα, γιατί Αυτά. Δεν μου επιτρέπουν να πάω παραπέρα. Και επειδή μας ενδιαφέρει τόσο πολύ το θέμα, θα κινηθούμε και γρήγορα, γιατί θέλουμε να κάνουμε κάποια βασικά πράγματα και από πλευράς χρονοδιαγράμματος. Ευχαριστώ και πάλι τους ε, ομιλητές για τις εξαιρετικές παρεμβάσεις, τον κύριο Νάση για την αναφορά και για όλη τη δουλειά που έχει κάνει για τους συναδέλφους από την Επιτροπή Αναφορών. Κάτι τελευταίο. Υπάρχουν θέματα ανθαγένειας, έχουμε την πολυπλοκότητα του ζητήματος, γιατί καλύπτουμε και αυτό το τομέα, αλλά και τόσους άλλους τομείς, ε, τα θέματα των ανηλίκων. Η πολυπλοκότητα όμως μόνο αυξάνει τη σημασία του ζητήματος και το ενδιαφέρον των μελών μας. Οπότε σας υπόσχομαι ότι θα δοθεί συνέχεια. Τα ξέρω πολύ καλά αυτά τα θέματα, γιατί όπως θα σας πει και η κυρία Ζωνόκα, έχω ασχοληθεί με αυτά εδώ και πολλά χρόνια και γνωρίζω τα συγκεκριμένα ζητήματα που θίγεται για τις μειονότητες και τα όσα συμβαίνουν. Ήθελα να το αναφέρω και αυτό. Και τέλος, Υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον και από πλευράς πολιτών. Αν δείτε και το έγγραφο, θα δείτε όλους τους φορείς που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια και τον αριθμό των πολιτών. Οπότε ευχαριστώ και όλους τους ε, αναδεικνύουν αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ για την ε, παρουσία σας. Ελπίζω να υπάρξει πραγματική συνέχεια και να δούμε αυτό το θέμα ε, με αυτή τη σύνθεση και με άλλες. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.